Mes Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σα. Κύριε Βαντενκάμ, πολλά καλά. Καλησπέρα σα, Πολύ ωραία. Ναι, ναι, ξεκινάμε. Είμαστε στην ώρα μας. Όχι, ξέρετε ότι στην Γαλλία προβλέπεται το ακαδημαϊκό τέταρτο. Λοιπόν, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Έχουμε το σχέδιο μερίσιας διάταξη. Μπορούμε να το εγκρίνουμε δεν υπάρχουν αντιρρήσει. Δεν βλέπω καμία αντίρρηση. Πολύ ωραία. Διάφορες συνακοινώσεις τώρα από την Πρόεδρο. Καταρχάς, να σας ενημερώσω για την τελευταία συνεδρίαση σε, σε, τους, ε, της διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών. Σα συγγνώμη, είναι Δευτέρα, όλοι ξεκινάμε, έκανε ε, ένα λάθος. Δεν πρόκειται τώρα να σα ενημερώσω για τη διάσκεψη των Πρόεδρων των Επιτροπών. Θα το κάνω αυτό κατά τη διάρκεια τη συνεδρίασης των συντονιστών. Σα το συγγνώμη. Περνάμε στα πρακτικά τη 31 ης Αυγούστου. Μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά. Δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. Ουδή. Πολύ ωραία. Ανακοινώσει τη Προέδρου. Πολύ απλά θα ήθελα να σα ξαναπώ ότι διοργανώνουμε την πρώτη εκδήλωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, μια εκδήλωση με τη συμμετοχή των πολιτών στις 11 Οκτωβρίου. Πρόκειται για μια τέτοια πρώτη εκδήλωση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτη φορά μια κοινοβουλευτική επιτροπή ανοίγει τι πόρτε στου Ευρωπαίου πολίτε για μια δημοκρατική συζήτηση όσον αφορά τι μεταφορέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλη λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μα παρακολουθήσει, καθότι θα μεταδοθεί η συνεδρίαση αυτή, η εκδήλωση αυτή μέσω των μέσων κοινωνική δικτύωση, μέσω του Twitter επίση. Ελπίζω λοιπόν να έρθετε πραγματικά στη συνεδρίαση αυτή και να είστε πολύ άριθμοι. Θα ήθελα επίση να μου και τους καλεσμένους σας πριν τις 26 του μηνός, δηλαδή μέχρι αύριο. Ο κύριος Μπάχνουμον παρακολουθεί νομίζω. Και μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης, ψηφοφορίες. Θα ήθελα να δοκιμάσουμε τώρα το σύστημα με τις κάρτες. Να δούμε αν έχουμε απαρτία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και όντως έχουμε απαρτία. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες πρώτη ψηφοφορία όσον αφορά την έκθεση για τη Διεθνή Διακυβέρνηση των Ωκεανών, πρώτη την έκθεση της κυρίας Μοντέιρο. Καλημέρα σας κύριε Μοντέιρο. Νιώθετε κάποια πίεση, σταχωμένη. Φοβάστε λιγάκι, όχι, όλα καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εγώ πρέπει να σου πω πραγματικά ότι είμαι σε φόρμα σήμερα, αισθάνομαι πολύ καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Συμβαστική παριθμό 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Βλέπω ότι είστε όλοι σε φόρμα. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Η τροπολογία 18 εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε τη τροπολογία 27. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κύριε Καπούτο, καλημέρα σας. Ψηφίζουμε τη δική σας τροπολογία. Τροπολογία 28 λοιπόν, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 61. Υπέρ. Κύριε Βαντεκάμπ, θέλετε επαλήθευση για τροπολογία 60, άρθρη ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Η τροπολογία 60, υπέρ 19, κατά 14 και εγκρίνεται. Τροπολογία 61, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 63. Η... Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 62. Πολύ ωραία. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. 63. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 73. Υπέρ παρακαλώ. Κατά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 Σύνολο τώρα του κειμένου, τελική ψηφοφορία, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. 31 υπέρ. Δύο αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Μοντέιρο. Η έκθεσή σας εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Ας συνεχίσουμε τώρα με την επόμενη ψηφοφορία. Και περνάμε στην επόμενη έκθεση που έχει να κάνει με την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρήση της κανονιστικής, διαδικασίας προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Μάιερ είναι ο εισηγητής, ο συντάκτης γνωμοδότησης. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα ψηφίσουμε καταρχάς τις τροπολογίες 44 έως 98. On block. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Το σύνολο αυτών τροπολογιών απορρίπτεται. Τροπολογία 99. Υπέρ παρακαλώ. Στην 99 είμαστε. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές η 99 εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα συνολικά τις τροπολογίες 1 έως 43. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Άρτε ψηφοφορία. Οι τροπολογίες 1 έως 43 εγκρίνονται. Περνάμε τώρα στις τροπολογίες 109 έως 7. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 111 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 112. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 113. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το τροπολογία 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα τις τροπολογίες 118 έως 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 120 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 121 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τελευταία τώρα τροπολογία, μάλλον συγγνώμη, τελική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, ενδεχομένως να κάνω λάθος, αλλά δεν ψηφίσαμε τις τροπολογίες 101 έως 106. Μέχρι την 98-99 φτάσαμε, αλλά νομίζω ότι δεν ψηφίσαμε εν συνεχεία τις τροπολογίες 100 έως 106 ή 101 έως 106, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό μου λένε και οι συνάδελφοι. Πρόεδρος, κύριε Γκολνίσο, όταν ψηφίσαμε από κοινού κάποιες τροπολογίες στο πρώτο, στο πρώτο σύλλογο, πήγα, στην πρώτη τροπολογίες πήγαμε από το 44 έως 99 και έπειτα καλύψαμε και αυτές τις οποίες αναφερθήκατε, 100-106. Έχουν εγκριθεί πάντως, ψηφίσαμε και έχουν εγκριθεί αυτές οι τροπολογίες. Λοιπόν, τελική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Η έκθεση συγκρίνεται λοιπόν με 22 ψήφους υπέρ και μία αποχή. Σας ευχαριστούμε πολύ και συνεχίζουμε με την μέρη διάταξη. Ολοκληρώσαμε τις προφορίες. Περνάμε στην ε, έκθεση για την επιτάχυνση της καινοτομία στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Βιομηχανίας. Συντάκτρα της γνωμοδότησης είναι η κυρία Ιζαμπέλα Ντεμόντε. Καλημέρα σας. Δώσω το λόγο, στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, στους και οδησηγητές καταρχάς και έπειτα σε οποιονδήποτε άλλο θέλει να πάρει το λόγο. Και εν τέλει θα καλέσω τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο και κυρία Συγήτρια θα σα ξαναδώσω το λόγο για να ολοκληρώσετε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η υφιστάμενη στρατηγική έχει ως στόχο να επιταχύνει την καινοτομία στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Η μετάβαση προς μία κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω μετά την έγκριση τη Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα. Εμεί ανέκαθεν καταβάλαμε πάρα πολλέ προσπάθειες και βρισκόμασταν στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, προωθώντας νέες πηγές ενέργεια και στη βιομηχανία και στι μεταφορέ και στα κτίρια. Η στρατηγική λοιπόν, προκειμένου να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, προβλέπει ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για τις ιδιωτικές επενδύσεις, να δημιουργηθούν δηλαδή κατάλληλες συνθήκες στην αγορά για να προωθηθεί η κοινοτομία. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στην κοινοτική χρηματοδότηση και στις νέες εκείνες τεχνολογίες, προκειμένου να καταφέρουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, με χαμηλή χρησιμοποίηση ορυκτών καυσίμων, καθώς επίσης και μεγαλύτερες δυνατότητες αποθήκευσης πλέον. Θα πρέπει να συνεργαστούν και τα κράτη-μέλη μεταξύ τους, αλλά και θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την καινοτομία και όσον αφορά την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή όπω προεβλέπεται από τη Συμφωνία των Παρισίων. Θα πρέπει όμω να επικεντρωθούμε και στον τομέα των μεταφορών. Ο τομέα αυτό ε, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βρισκόταν ε, εκτό του συστήματο εκείνου που προβλέπει μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ξεκινώντα λοιπόν από μια βιώσιμη αστική κινητικότητα και επομένω πιο αποτελεσματική, φτάνοντας σε πιο αυτόνομα συνδεδεμένα οχήματα, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και υποστήριξη στις κοινοτομίε εκείνες που προωθούν τις ε, βιώσιμες καθαρές μορφές ενέργειας και μειώνουν την ηχορύπανση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικεντρωθούν ε, οι προσπάθειέ μα στη δημιουργία ευφυών διαθεσιστεδεμένων πόλεων μέσω συγκεκριμένων στόχων βιωσιμότητο, μέσω στόχων ασφαλεία των οδικών μεταφορών και προστασία τη δημόσια υγεία. Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα στον τομέα του τουρισμού. Βλέπουμε όλο και περισσότερο ότι φτάνουν όλο και περισσότεροι τουρίστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό προφανώ από μόνο του είναι πάρα πολύ θετικό. Η πρόσβαση όμω στι δημόσιε μεταφορέ από του τουρίστε είναι πάρα πολύ χαμηλή ακόμα. Είναι πάρα σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε μέσω των καθαρών μορφών ενέργειας και μέσω πιο βιώσιμων, μεταφορών να καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερα κίνητρα προκειμένου τουρίστες να χρησιμοποιούν περισσότερο τις δημόσιες μεταφορές. Ελπίζω ότι ο σημαντικότερος αυτός τομέας των μεταφορών αλλά και του τουρισμού θα καταφέρει να δραματίσει στο μέλλον ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την κοινοτομία για τις καθαρές μορφές ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να ξεκινήσει τώρα η συζήτηση και δίνω ευθύ αμέσω το λόγο στην κυρία Κλούνε. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και την εισηγήτρια για τη συνεισφορά της. Η αποτελεσματική δράση στον τομέα της ε, ενέργειας είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η παραγωγή ενέργειας ευθύνεται για το 80% των εκπομπών που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η πρωτοβουλία αυτή λοιπόν είναι πολύ ευπρόσδεκτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να επιταχύνουμε την καθαρή ενέργεια και η Επιτροπή μας θα έχει την ευκαιρία να συμβάλλει στην έκθεση και να δώσει τη γνώμη της. Η κλιματική αλλαγή είναι πρόβλημα για εμάς. Πρέπει να αναλάβουμε γρήγορη δράση για να το λύσουμε και να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα. Αυτό είναι ευκαιρία για την Ευρώπη, ενισχύει την ευημερία των πολιτών, βελτιώνει την ποιότητα του αέρα, ανοίγει νέε πόρτες, δίνει νέε ευκαιρίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος παγκοσμίως στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, στις μεταφορές, στα κτίρια, στις υποδομές κτλ. Όμως ε, σε κάποια πράγματα υστερούμε. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, δεν είναι και πολύ ανταγωνιστικές από άποψη κόστους θα πρέπει να υιοθετηθούν ταχύτερα τα υφιστάμενα αποθέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και να κάνουμε το πάνω έτσι ώστε οι πόλεις και οι περιφέρειες να είναι καλά εξοπλισμένες, να ενισχύσουμε την ε, επένδυση και να αναπτύξουμε καθαρές μορφές ενέργειας το συντομότερο δυνατόν. Θα ενθαρρύνουμε έτσι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα προωθήσουμε τη βιώσιμη χρηματοδότηση όλων των εταίρων για να συνεχίσουν οι επενδύσεις και η καινοτομία στον τομέα αυτό. Η καινοτομία είναι ένα από τα βασικά και πρέπει να δώσουμε έμφαση και να το τονίσουμε αυτό στην έκθεση. με το θεματολόγιο αυτό για την καλύτερη τοποθέτηση και τους καλύτερους κανονισμούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα των νέων προτάσεων και εδώ μπορούμε να παρέμβουμε. Τα συστήματα μεταφορών έχουν πάρα πολλές δυνατότητε, αλλά είναι και μεγάλη πρόκληση για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποστηρίξουμε τις έξυπνες υπηρεσίες κινητικότητας περισσότερη καινοτομία χρειαζόμαστε στον ηλεκτρισμό νέας γενιάς, στα ηλεκτρικά κινούμενα αυτοκίνητα, με μπαταρίες που θα ε, δίνουν μεγαλύτερη αυτονομία, με μεγαλύτερη διάρκεια και που θα ενισχύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Πρέπει να έχουμε καινοτομία και στις υποδομές. Αυτή είναι η λέξη κλειδί. Να κάνουμε τα παν για να συμβεί για να έχουμε μια οικονομία με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα. Και βεβαίως χρειαζόμαστε νέες ψηφιακέ τεχνολογίες για νέα ολοκληρωμένα ενοποιημένα συστήματα αστικών μεταφορών. Θα συμβάλλουμε για τη σύνταξη του κειμένου προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Φώστερ για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Θέλετε το λόγο? Όχι καλός. Ο κύριος Τελίνσκα από τους φιλελεύθερους, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα, συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του αρμοδίου συναδέλφου, του οποίου η πτήση καθυστέρησε. Αυτό είναι το μειονέκτημα των βουλευτών που έρχονται από απομακρυσμένε περιοχές και μου ζήτησε να του παρουσιάσω τι, απόψεις τους, τις απόψεις του για το θέμα που μας απασχολεί. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ντεμόντε για την πολύ καλή γνωμοδότηση, για, τη σημασία που, για το πόσο σωστά απεικόνισε τη σημασία που έχει ο τομέα των μεταφορών στη μεταβατική αυτή περίοδο προ μια οικονομία με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα. Καλωσορίζουμε την ε, θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πιο καθαρέ υποδομέ και για εναλλακτικέ της ε, λύσεις μεταφορών. Η νέα προσέγγιση διασυνδέει την ενέργεια, τι μεταφορέ και τι ψηφιακέ τεχνολογίε και εκτιμούμε ιδιαίτερα σε αυτή τη νέα προσέγγιση που έχει οθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σκεπτικό της. Οι ορεινέ περιοχές, οι εξόχως απόκεντρες, οι απομακρυσμένες, οι περιοχές της υπαίθρου δεν αναφέρονται στην έκθεση και αυτό οφείλουμε να το τονίσουμε. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την υφιστάμενη χρηματοδότηση, να την εστιάσει και να την επικεντρώσει με πιο συγκεκριμένο τρόπο σε συγκεκριμένες προτεραιότητες, όπως η ηλεκτροκινητικότητα και η ενοποίηση των συστημάτων μεταφορών εντός του άστεως αλλά και εντός της υπαίθρου, έτσι ώστε κανείς να μην μείνει πίσω. Χαιρόμαστε διότι υπάρχει αυτό το θεματολόγιο με τους ε, οδικούς χάρτες και αντίστοιχους κυβερνητικούς μηχανισμούς και μηχανισμούς διακυβέρνησης και διαχείρισης για να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί οι επενδύσεις, η καινοτομία. Όλα αυτά τα προγράμματα και τα έργα είναι πολύ σωστά και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Ήπεθρο και στις δυνατότητές της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει τις προτάσεις της, δεν έχει μια λύση μία και μόνο που να ταιριάζει, σε όλες τις περιπτώσεις. Αντιθέτως, μιλάμε για μεταβλητή ε, γεωμετρία αναλόγως με την ε, κάστοτε περιφέρεια και τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της. Για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής στην Ήπεθρο πρέπει να έχουμε τα καλύτερα προσόντα, τις καλύτερες δεξιότητες, τις καλύτερες και βέλτιστες λύσεις οι οποίες να κυκλοφορήσουν και να διαδοθούν. Τέλος, να πω ότι ο μόνος τρόπος να παραμείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο είναι να τους δίδονται ευκαιρίες, να μπορούν να βρουν δουλειέ, να έχουν καλές μεταφορικές συνδέσεις με την πρωτεύουσα, να, έχουν, να υπάρχει σωστή ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και να έχουμε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας και στην Ήπεθρο. Αυτά έχω να σας πω εξ ονόματος του αρμοδίου συναδέλφου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Κράμερ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και προς την συντάκτρια. Ε, ο δικός μας ε, σκιώδης συγητής, ο Μπάσεκ Χαουτ, λείπει. Θέλω να πω το εξής. Στις πόλεις ε, η κυκλοφορία η οδική ευθύνεται κατά 70% για τις, τους παγκόσμιους ρήπους. Για να αλλάξει κλιματική αλλαγή που πρέπει να αλλάξει και θέλουμε να την τερματίσουμε, συμφωνούμε όλοι στα λόγια αλλά στα έργα λιγότερο. Πρέπει να αλλάξει η κατάσταση λοιπόν τη κυκλοφορία στους πόλεις. Ε, στις 5 Οκτωβρίου του 2015 συμφώνησαν με όλοι οι Υπουργοί Μεταφορών ε, να ε, μετατοπιστούν οι μισές μεταφορές της πόλης, εμπορικές μεταφορές, Παρίσι, Λονδίνο, Μαδρίτη, να φύγει από τα φορτηγά και να πάει στην ηλεκτροκίνηση παραμένει η δυνατότητα ε, προμηθειών φορτίων, αλλά χωρίς φορτηγά. Αυτά είναι ποδήλατα ε, επίσης που λέγονται cargo bikes. Ε, είναι ποδήλατα που μπορούν να μεταφέρουν φορτία και οι πόλεις παραμένουν καθαρές. Δυστυχώς η Γερμανία εδώ είναι αρνητικό παράδειγμα. Ξέρουμε ότι τα στοιχεία που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν τηρούνται, δεν γίνεται να τηρούνται στις περισσότερες πόλεις μας. Αν αντικαταστήσουμε όμως τα φορτηγά για τις προμήθειες των καταστημάτων από τα λεγόμενα ε, φορτηγά ποδήλατα, cargo bikes, ε, τότε θα σωθούμε. Όταν μιλάμε για την ηλεκτροκίνηση, ε, γίνεται λόγος κατά 95% για τα ε, αυτοκίνητα, Να υπάρχουν και ποδήλατα. Ο Φόγγελ, ε, δήμαρχος του Μονάχου πριν από 45 χρόνια, ζει ακόμα ο άνθρωπος, είπε ότι το αυτοκίνητο είναι ο θάνατος για τα κέντρα των πόλεων μας. θα συνεχιστεί ε, ο θάνατος των πόλεων και η δολοφονία ακόμα και αν αντικαταστήσουμε τα αυτοκίνητα και με ανανεώσιμες που δεν γίνεται αυτό αύριο. Λοιπόν, θα πρέπει να μειώσουμε και τον αριθμό των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην πόλη. Κάποιος επίσης είπε ε, παλιά ένας Γερμανός Υπουργός Μεταφορών ότι το 90% ε, των μετακινήσεων στις πόλεις με αυτοκινήτα είναι μικρότερο των 6 χιλιόμετρων. Λοιπόν, να μην κοιτάμε μόνο ε, τα προ... Να δείτε τι γίνεται με το τρένο. Μας λείπουν 25 ε, χρόνια για να ε, κλείσουμε τα προβλήματα ηλεκτροκίνησης που έχει το τρένο, ας πούμε από το Βερολίνο για να πάει στο Βρότσλαβ, 300 χιλιόμετρα, έχουμε μηχανή, δίζελ τρένο και λείπουν 50 χιλιόμετρα ε, για να ηλεκτροδοτηθούν και δεν μπορούμε. Περιμένουμε 25 χρόνια. Ενώ δίνουμε χοντρά λεφτά για τα αυτοκίνητα και στη Γερμανία προωθούν το αυτοκίνητο και του αυτοκινητοδρόμου. Θα πρέπει να βλέπουμε λοιπόν ποια ε, προγράμματα έχουν συγχρηματοδότηση, πώ πιάνουν τόπο τα χρήματά μα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει να το προωθεί. Να μην ε, κοιτάει τι θέλουν τα κράτη μόνο, αλλά να επενδύουμε και στην ηλεκτροκίνηση. ο κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Ιζαμπέλα για την εργασία που έχει κάνει για το ζήτημα αυτό. Είναι πραγματικά πολύ καλή η εργασία της και το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό γιατί αναφερόμαστε εδώ στον τομέα της κοινοτομία όσον αφορά την καθαρή ενέργεια. Εδώ μιλάμε πραγματικά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα πρέπει να διαμορφωθεί με χαμηλές εκπομπές του οξύδου του άνθρακα και εμείς ως Επιτροπή βρισκόμαστε πραγματικά στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα. Η κοινοτομία και η τόνωσή της δεν μπορεί να περνάει μόνο μέσω τη έρευνας γιατί Ουσιαστικά εδώ έχουν καταβληθεί πολύ σημαντικέ προσπάθειε τελευταία χρόνια, μην το ξεχνάμε αυτό. Πρέπει όμω παράλληλα να δοθεί και μία όθηση από τον ίδιο το βιομηχανικό κλάδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να δημιουργηθούν οι απαραίτητε συνέργειε μεταξύ έρευνα και παραγωγικού κλάδου, προκειμένου να υλοποιηθεί στην πράξη η νέα αυτή επανάσταση που θέλουμε στο βιομηχανικό τομέα. Ξέρετε ότι η μετάβαση αυτή προς την βιωσιμότητα αποτελεί πραγματικότητα σε άλλες περιοχές του κόσμου που έχουν δημιουργηθεί και σχετικές θέσεις απασχόλησης. Μάλλον υπολοιπόμεθα λίγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και μάλλον πρέπει να καταβάλουμε λίγες περισσότερες προσπάθειες, ιδίω όσον αφορά τον τομέα των εφιών μεταφορών. Ακριβώς λοιπόν στον τομέα αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθούν περισσότεροι χρηματοδοτικοί πόροι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα πρέπει καταρχάς να υποστηρίξει κυρίως χρηματοδοτικά τον κλάδο αυτό προκειμένου να κινητοποιηθούν και περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, απευθύνομαι τώρα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος θέλει το λόγο. Α, κύριε Γκολνίσσα, δεν σας είχα δει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν θα με ακρηγορήσω. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όσο και σημαντικό το θέμα μας. Να επιμείνω μόνο λίγο στο εξή σημείο που θεωρώ ότι θα το εξετάσει η συγγήτριά μας. Τις περισσότερες φορές, για να αποφύγουμε ε, την, ε, ε, ε την κίνηση στις πόλεις ε, Ανατρέχουμε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θέλω να σας πω όμως ότι ο ηλεκτρισμός όπως όλοι γνωρίζουμε ή θα πρέπει να γνωρίζουμε δεν είναι πηγή ενέργειας, είναι μόνο φορέας ενέργειας. Δηλαδή το ρεύμα πρέπει να το παράγει κάποιος από κάπου. Οπότε ε, είτε αυτό γίνεται ε, σε θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, οπότε ε, δεν είναι θετική η το ισοζύγιο ε, του διοξιδίου του άνθρακα, είτε παράγεται από την πυρηνική ενέργεια κυρίως, σε πυρηνικά εργοστάσια, όπου εδώ έχουμε άλλα προβλήματα και αντιστάσεις δεδομένης ε, της ε, επικενδυνότητας αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας, της παραγωγής της πυρηνικής. Θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Εγώ, ξέρετε, ζω στο Παρίσι και φυσικά ενδιαφέρομαι για κάθε μέτρο που μπορεί να καταστήσει την κυκλοφορία πιο ρευστή και να μην έχουμε ε, κυκλοφοριακή συμφόρηση, ποτηλιαρίσματα, όπου προκαλείται ρήπαση του περιβάλλοντος, εκνευρισμός του πληθυσμού, ε, καθυστερήσεις κτλ. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Je... Και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα σας δώσω το λόγο. Είναι αρκετά σημαντικό να διαβάζουμε τον τίτλο γιατί πρόκειται για την καινοτομία, για μια καθαρή ενέργεια. Δεν έχουμε 100.000 ε, καθαρές ενέργειες. Έχουμε την αιωλική, την ηλιακή. Αυτές είναι καθαρές ενέργειες που δεν ε, εκπέμπουν ε, Τώρα στην Ευρώπη όλοι θέλουν να στραφούν το, στο περίφημο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αλλά ε, σήμερα οι παραγωγοί, οι κατασκευαστές δεν είναι έτοιμοι. Σήμερα δεν είναι έτοιμοι οι εργαζόμενοι, δεν είναι κατευθυσμένοι και αύριο δεν θα έχουμε μόνο την ηλεκτρική ενέργεια, θα έχουμε και άλλες μορφές. Το υδρογόνο, το αέριο. Ε, ενεργειακό μείγμα που θα προχωρήσει ως τεχνολογία. Και προσοχή, γιατί Αύριο θα συζητήσουμε για το μέλλον των μεταφορών. Αλλά το αυριανό αυτοκίνητο δεν θα είναι μόνο πιο καθαρό, θα είναι και ένα αυτοκίνητο που θα μοιραζόμαστε με άλλους. Και όταν μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε και για αυτόνομη οδήγηση. Άρα, όλες αυτές είναι ρηξικέλευθες αλλαγές και πολύ συναρπαστικές, αλλά έχετε δίκιο κύριε Καπούτου, θα πρέπει να γίνεται λόγος για πραγματικές επενδύσεις. Γιατί αν δεν επενδύσουμε σήμερα εκεί, ουσιαστικά στην καινοτομία, σε καμία περίπτωση δεν προετοιμάζουμε το μέλλον, πόσο μάλλον τις μελλοντικές γενιές που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους και την κατάσταση του πλανήτη, αλλά και ε, μια τελείως νέα κινητικότητα, με νέα δεδομένα. Μετά από αυτά τα εισαγωγικά, θα δώσω το λόγο στον κύριο Κουινάγα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστεί την κυρία Ισαπέλα Τελμόντε για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης για την καθαρή ενέργεια και την καινοτομία. Οι υποδείξεις και οι προτάσεις στηρίζουν την ε, πρωτοβουλία για την πολιτική, θα βοηθήσουν πολύ για την εφαρμογή του, της ανακοίνωσης, του ανακοινωθέντος το να βελτιώσουμε την πρόσβαση των πολιτών σε λύσεις με χαμελό ενεργειακό αποτύπωμα είναι στο επίκεντρο των φιλοδοξιών μας και ημών και των πολιτών. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για την επιτάχυνση της καινοτομίας. Προηγμένες λύσεις αποθήκευσης, προηγμένες ε, υποδομές, υπηρεσίες έξυπνης κινητικότητας είναι βασική προτεραιότητα, όχι μόνο για να επιταχύνουμε την έλευση της καθαρής ενέργειας, αλλά και για να ενισχύσουμε αυτή το ε, θεματολόγιο που υιοθετήθηκε το Μάιο του 2017 για τις μεταφορές και την ενέργεια. Και θα συνεχίσουμε να το στηρίζουμε μέσα από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Η ανάγκη και η πρόκληση να ε, έχουμε κοινοτομίες τις οποίες να ανεβάσουμε σε υψηλότερα επίπεδα και να τις απλώσουμε, να τις διαδώσουμε σε περισσότερα ακροατήρια είναι απαραίτητη. Είναι κάτι το απαραίτητο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει την ηλεκτροκινητικότητα και τις ολοκληρωμένες και ενοποιημένες αστικές μεταφορές. Οι συγκεκριμένες δράσεις προβλέπονται, εκτός από τις πρωτοβουλίες μας, προβλέπονται και στον ορίζοντα 2020 και αλλού. Και έχουμε οδικούς χάρτες και είναι πρωτοβουλίες ανοιχτές που απευθύνονται και στην Ήπεθρο. Με την ε, διαχείριση αυτή ε, ενοποιημένη διαχείριση μεταφορών και ενέργειας θα έχουμε νέα προσέγγιση για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και πολύ καλύτερες λύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Η κυρία Ντεμόντε παρακαλώ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδης ηγητές και όλους τους συναδέλφους αλλά και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις παρεμβάσεις τους. Πραγματικά τα όσα έθιξαν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, να δημιουργηθεί όντως ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο με τη δημιουργία και την προώθηση επενδύσεων για την καθαρή ενέργεια. Το είπα αυτό και στην αρχική μου έκθεση, στην αρχική μου παρέμβαση. Μόνο μέσω των επενδύσεων αυτό θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση και εν τέλει θα καταφέρουμε να ελοποιήσουμε την ευκταία αυτή κοινοτομία. Νομίζω όμω ότι θα πρέπει να έχουμε και μια νέα προσέγγιση, ένα σύστημα bottom-up, από την βάση προ την κορυφή, όπου δεν θα δραστηριοποιούνται μόνο οι μεγάλε επιχειρήσει, αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολλές φορές και οι ο ο όσον αφορά την ψηφιοποίηση και αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να έχουμε και νέους ψηφιακούς φορείς και μπορούμε όντως στο μέλλον να μοιραζόμαστε όλο και περισσότερο, για παράδειγμα τα οχήματα όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε. Αυτό δεν αποτελεί μόνο χαρακτηριστικό του μέλλοντος αλλά συμβαίνει όντως και στο παρόν και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπε και οι συνάδελφοι, να επενδύσουμε περισσότερο σε πιο απομακρυσμένες περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην Ήπεθρο. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε διασυνδεδεμένες υπηρεσίες, δυνατότητες μεταφοράς και για τις περιοχές αυτές, προκειμένου τελικά να μην φεύγει από εκεί πέρα ο πληθυσμός. Ο κ. Κάμερεν συνεχεία αναφέρθηκε στις πόλεις εκείνες, οι οποίες, στις οποίες θα πρέπει να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση, όχι μόνο για τις μεταφορές των εμπορευμάτων, αλλά και για τις μεταφορές των επιβατών. Και να ολοκληρώσω τέλος λέγοντας ότι πιστεύω και εγώ ότι θα πρέπει να γίνουν πράγματι επενδύσεις και μέσω του ΕΦΣΥ και χρησιμοποιώντας έτσι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι η καθαρή ενέργεια δεν είναι μόνο κάτι το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτόνομα, αλλά και κάτι το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να δημιουργήσουμε άλλε μορφέ ενέργεια, όπω για παράδειγμα την ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια δεν παράγεται μόνο από τα ορυκτά καύσιμα, έτσι δεν είναι. Τούτων λεχθένω θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ντεμόντε. Θυμίζω την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 4 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Και συνεχίζουμε. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Διάσωση ζώων, ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δική σας έκθεση κύριε Κόχιν αυτή, έκθεση προτεραιότητας. Είναι απίστευτα τα στοιχεία. 120.000 ζωές χάνονται κάθε χρόνο δυστυχώς στην άσφαλτο 120.000 ανθρώπινες τραγωδίες. Γιατί για κάθε νεκρό από τροχαίο έχουμε 7 τραυματίες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Η έκθεση είναι έκθεση προτεραιότητας για την Επιτροπή μας. Έχετε το λόγο κύριε Κόχ και στη συνέχεια οι σκιώδεις ηγητές και πάει λέγοντας. Θα ρωτήσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, εισηγητής. Ja, vielen Dank, Frau Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την ευγενική σας εισαγωγή. Αγαπητοί συνάδελφοι, την περασμένη εβδομάδα σε μία μέρα ε, τρία φορτηγά έπεσαν ε, σε ποτηλιάρισμα χωρίς φρένα, χωρίς να φρενάρουν, με ένα θύμα. Και το Σάββατο, πολύ κοντά στη γειτονιά μου, τη νύχτα, ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο, δεραπάρισε, ε, ο άνθρωπος ο οδηγός ε, εκτινάχθηκε και έχασε τη ζωή του. Εάν ε, φορούσε ζώνη, θα ζούσε ο οδηγός και αν είχε ένα σύστημα υποβοήθησης οδήγησης, επίσης θα είχε αποτραπεί το ατύχημα, το δυστύχημα μάλλον. Ε, θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν του συναδέλφους. Είναι σημαντική η έκθεση αυτή. Έχουν γίνει σημαντικές τροπολογίες ε, και πάρα πολύ χρήσιμες συμπληρώσει. Και με μεγάλη χαρά να τα συμπεριλάβω σε συμβαστικέ προτάσεις, αν δεν το έχω ήδη κάνει. Συνολικά είναι 226 οι τροπολογίες που κατατέθηκαν, 77 από το ΕΛΚ, 52 από τους σοσιαλδημοκράτες, 31 από τους φιλελευθέρους, 10 ECR, 20 των Πρασίνων, 23 από τη Γοέ και 13 από την ΕΝΕΦ. Προσωπικά έχω καταθέσει 16 τροπολογίες ε, γιατί υπήρχαν ανακρίβειες στη μετάφραση από τα γερμανικά στα αγγλικά. Δυστυχώς αυτά που λένε τα ρουμανικά τώρα δεν μπορώ να τα καταλάβω. Παράδειγμα, στην αρχική μου γερμανική έκδοση ε, ε, μιλώ για ένα σύστημα που στα αγγλικά το λένε departure warning. Δεν είναι αυτό. Το departure warning σε ειδοποιεί ότι έχεις φύγει από την λωρίδα σου, ενώ το άλλο σύστημα επεμβαίνει ε, μαλακά για να σε κρατήσει στην ίδια λωρίδα. Γενικά, ε, θα κάνω 32 συμβαστικές που καλύπτουν 145 τροπολογίες, περισσότερες από τις μισές όλων όσες έχουν κατατεθεί. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Ήταν εξαιρετικές οι ιδέες πάρα πολλών συναδέλφων και δεν μπορώ παρά να τις υποστηρίξω και να συστήσω να υπερψηφιστούν. Συγκεκριμένα, πρώτον, υπάρχει μεγάλη συναντήληψη και ομοψυχία για τους ανθρώπους που έχουν αναπηρίες, που έχουν προβλήματα στην κινητικότητα, χρειάζεται ιδιαίτερη μέρημνα και προσοχή για αυτού. Αυτό αφορά κυρίω τον τρόπο με τον οποίο ε, ε, ε ακούν τα προειδοποιητικά ε, σήματα και σε ε, ποια ένταση του ήχου. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στατιστικά στοιχεία αξιόπιστα έτσι ώστε να αποφύγουμε μελλοντικά δυστυχήματα. Από την άλλη τα στοιχεία αυτά βεβαίως θα πρέπει να παραμένουν ανώνυμα και να έχουν και περιορισμούς στη χρήση και τη διάδοσή τους. Στη συνέχεια. Στα μεγάλα φορτηγά υπάρχουν τυφλές και νεκρές γωνίες που πολλές φορές ε, τους εμποδίζουν να βλέπουν την κίνηση και την κυκλοφορία. Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες που δυστυχώς δεν μπορώ να τις ε, υποστηρίξω και να τις εγκρίνω, αλλά σας ευχαριστώ για αυτές γιατί είναι τροφή για σκέψη. Ε, σε μία τροπολογία ε, να σας πω γιατί την απορρίπτω, είπα πάση δεν την λαμβάνω υπόψη. Αυτή είναι έκθεση πρωτοβουλία και δεν έχουν μεγάλη θέση κάποιε τροπολογίε, γι' αυτό τι έχω απορρίψει. Ή θέλουν να στρέψουν την έκθεση σε μια τελείω διαφορετική νέα κατεύθυνση ε, ή ε, κάποια άλλα θέματα που τα θεωρώ τελείω περιτά σε μια έκθεση πρωτοβουλία. Κατέληξα λοιπόν κατόπιν ορίμου σκέψεως να προτείνω να απορριφθούν, να μην ληφθούν υπόψη τροπολογίε ή τμήματα τροπολογιών που αναφέρονται σε αίτια αναφοράς. Μέχρι πότε ποιο σύστημα υποβοήθησης οδήγηση θα πρέπει να έχει υιοθετηθεί, αυτό συνειδητά το απέφυγα στην έκθεση μου. Υπάρχουν συνάδελφοι που προτείνουν συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, ε, που ε, επιτρέψτε μου να πω θεωρώ ότι έχει επιλεγεί αυθαίρετα. Παρακαλώ να μην με παρεξηγήσετε. Και εγώ ε, θέλω να υπάρχουν στόχοι φιλόδοξοι και προθεσμίες φιλόδοξες. Ωστόσο, τόσο συγκεκριμένες απαιτήσει δεν θα πρέπει να τις βάζουμε σε έκθεση πρωτοβουλία. Από εκεί και πέρα θα ήταν και ασυνεπές να βάλουμε προθεσμία για κάποια συστήματα τα οποία θεωρούμε πάρα πολύ απαραίτητα και ε, αναγκαία, ενώ για κάποια άλλα όχι. Γιατί τελικά στην αγορά κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή ε, διάφορα συστήματα ασφαλείας. Από την άλλη υπάρχουν και επιχειρήματα πολύ πιο έγκυρα. Θα πρέπει να πιέσουμε να περάσει ο κανονισμός για τη γενική ασφάλεια των οχημάτων στην αρχή του 2018. Και εκεί λοιπόν είναι ε, το σωστό σημείο και όχι μια έκθεση πρωτοβουλία να αναφέρουμε προθεσμίες για την ε, γενίκευση της χρήσης αυτών των μηχανισμών. Και σε περίπτωση που δεν μας φανούν αρκετά φιλόδοξα αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ζητήσουμε συγκεκριμένες αλλαγές, αλλά σε συγκεκριμένα άρθρα ή παραρτήματα. Η σημερινή έκθεση, επαναλαμβάνω, έκθεση πρωτοβουλίας και θα πρέπει να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να συμφωνήσουμε τι συστήματα ε, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά στα νέα τα ε, στα, στις σειρές των ε, μοντέλων. Επίσης, στο στάνταρ εξοπλισμό. Κάποιες άλλες τροπολογίες ε, θέλουν να προτείνουν κίνητρα και μόνο. Αυτό είναι πάρα πολύ χαλαρή ε, πρόταση και μεγάλη επιστοδρόμηση Κατά την ψήμη χάνουμε και τον πραγματικό μας στόχο, που είναι η ε, αύξηση της οδικής ασφάλειας. Κάποιες άλλες τροπολογίες αφορούν τη δυνατότητα να αγνοεί κανείς, να αποσυνδέει ή να σβήνει όλα αυτά τα συστήματα. Ορισμένοι συνάδελφοι θέλουν να μην ε, ε, σηκώνουν καμία παρέμβαση ή καμία ε, κίνηση από πλευράς του οδηγού που θα τα καταργεί. Άλλοι δεν θέλουν καθόλου να συμβαίνει αυτό. Συγκεκριμένα, θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο γενικά να απαγορεύεται να επέμβει ο οδηγός για να καταργήσει το σύστημα. Καμιά φορά ε, ο οδηγός ε, θέλει να κάνει μια μανούβρα, έναν ελιγμό για να, για να μην τρακάρει. Δεν μπορεί να τον επαναφέρει στη λωρίδα το, το σύστημα υποποίησης. Μπορεί ε, να υπάρχει λόγος να αγνοήσει αυτό το σύστημα λόγω κακής και μια ασφαλούς οδήγησης ε, κάποιων άλλων οδηγών ή αν έχει φρένο ε, η κόφτη στα χιλιόμετρα μπορεί να χρειαστεί να επιταχύνει παρά το γεγονός ότι απαγορεύεται αυτή η ταχύτητα στη συγκεκριμένη ε, οδό για να αποφύγει ατύχημα. Δεν είναι δυνατόν να μην επιδέχεται καμία παρέμβαση το σύστημα. Μετά, δεν υπάρχει γενική λύση σε αυτό που προτείνει. Υπάρχουν συστήματα που βοήθησης οδήγησης, όπως είναι, ας πούμε, η πέδηση δεν θα πρέπει να μπορεί να διακόπτεται γιατί μπορεί να ξεχάσει ο οδηγός να το ενεργοποιήσει ξανά. Ή άλλα συστήματα όπως είναι το ηλεκτρονικό τηλεφώνημα ή το σύστημα αυτό που σε κρατάει στην ίδια λωρίδα ε, θα μπορούσε να διακόπτεται. Ε, για κάποια άλλα συστήματα που εξυπηρετούν μόνο την άνεση της οδήγησης και όχι την ασφάλεια, δεν υπάρχει πρόβλημα ε, να μπορούν να απενεργοποιούνται. Για μένα θα πρέπει αυτό να γίνεται σε δύο στάδια. Να μπορεί σε πρώτη φάση ο οδηγός να απενεργοποιεί το συναγερμό που χτυπάει, γιατί αυτό είναι το εκνευριστικό. Και σε δεύτερη φάση το ίδιο το σύστημα. Ε, και μετά όμως κάθε φορά που βάζει μπρος τον κινητήρα να επανέρχεται στην πλήρη λειτουργία το σύστημα βοήθησης. Τώρα, αν θα είναι αυτό αυτόματο, ε, μετά από κάποια ε, χρονική περίοδο θέλω να το συζητήσω με τους κοιότητες ηγητές και ίσως να μιλήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Αύριο το απόγευμα θα συνεδριάσουμε για πρώτη φορά με τους κοιότητες ηγητές για να συζητήσουμε τις 32 συμβαστικές μου τροπολογίες που έχουν στα χέρια τους οι σκιώδεις εδώ και λίγες μέρες. Η ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή μας έχει προβλεφθεί για τις 12 Οκτωβρίου και στο τελικό αποτέλεσμα θα συμμεληφθούν και οι προτάσεις της ε, Επιτροπής ΙΜΚΟ εσωτερική Αγοράς και ε, Προστασίας των Καταναλωτών, η οποία γνωμοδοτεί. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Περιμένω τις προτάσεις σας και σας ευχαριστώ για τις καταπληκτικές τροπολογίες που έχετε υποβάλει. Ευχαριστώ. Merci. Σας ευχαριστώ. Να δώσω το, το λόγο στην κυρία Σενάλοβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοχ, τον ε, εισηγητή για τις συμβαστικές προτάσεις του. Είπε ότι αύριο έχουμε την πρώτη συνεδρίαση των σχεδόν εισηγητών, άρα η σημερινή συζήτηση γίνεται πριν συνεδριάσουν οι σκιώδεις. Τώρα αρχίζει η συζήτηση. Στόχος αυτής της έκθεσης ποιος είναι. Η οδική ασφάλεια. Και η βελτίωση της ασφάλειας των οχημάτων. Όταν όμως συζητούμε οδική ασφάλεια, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την ασφάλεια των οχημάτων, αλλά και με την ασφάλεια των υποδομών, των αυτοκινητοδρόμων και άλλων. Αυτό ε, το έχω αναφέρει σε πολλές από τις τροπολογίες μου και ελπίζω να ληφθεί υπόψη στην τελική εκδοχή του κειμένου. Έχουμε δει ήδη τις συμβαστικές προτάσεις και φυσικά τις περισσότερες μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Για παράδειγμα, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε ειδικέ ομάδε, κινδύνου, ε, να έχουμε έλεγχο τη ταχύτητας ή κάποια άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν όχι με την ενεργητική αλλά με την παθητική ασφάλεια ε, που να λαμβάνει υπόψη περισσότερο τους ποδηλάτες και τους πεζούς. Ε, στις λεπτομέρειες θα τα συζητήσουμε και βεβαίως είμαστε υπέρ μιας συμβαστικής λύσης. Και τέλος, να αναφέρω ένα ακόμα θέμα. Να υπάρξει εναρμόνιση ε, των τιμών κατανάλωση ενοπνεύματος. Λέτε, υπάρχουν χώρες που είναι πάρα πολύ αυστηρές, δεν θα πρέπει να χαλαρώσουν, δεν πρέπει να είναι μια εναρμόνιση προς τα κάτω για τη συγκέντρωση συνοπνεύματος των οδηγών και της επιτρεπόμενης συγκεντρώσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιωτόσκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Κόχ. Είναι πολλές οι τροπολογίες και με τις περισσότερες συμφωνούμε λέει ο κύριος Λοτόφσκι. Στηρίζουμε την προσέγγιση του εισηγητή, αλλά έχουμε υποβάλει και τις δικές μας τροπολογίες, την 7 και την 104. Είναι πολύ σημαντικές, γιατί μιλούν για την αναγκαιότητα να βελτιωθεί η ασφάλεια των χρηστών του δρόμου και βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Ξέρετε, στην Πολωνία ο στόλος των αυτοκινήτων ήταν, είναι αρκετά παλιός και θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος μέχρι να εγκατασταθούν τα συστήματα που συζητείτε στην έκθεσή σας και αυτό θα σημαίνει πάρα πολλά θύματα. Έχουμε καλές τεχνολογίες που βελτιώνουν την ασφάλεια και θα πρέπει να προωθήσουμε αυτές τις λύσεις και να ενθαρρύνουμε τους ασφαλιστές και τους κατασκευαστές αυτοκινήτων τις αυτοκινητοβιομηχανίας να δώσουν κίνητρα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο σε ό,τι αφορά την ένταξη νέων συστημάτων στα οχήματα είναι η υψηλή του τιμή. Άρα και η αυτοκινητοβιομηχανία θα πρέπει να έχει τιμολογιακές πολιτικές φιλικές προς το καταναλωτή και το ίδιο ισχύει και για τα ηλεκτρικά οχήματα παρεμφερείς λύσεις, πιστεύουμε, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εδώ, γιατί η ζωή του ανθρώπου, η ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη υγεία είναι τόσο σημαντικά όσο και η προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριος Βαν Μίλτεμπορκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Συμφωνώ. Ε, εγώ Βέβαια μιλώ τώρα ε, εξ ονόματος του Γιένς Ρόντε, δεν θα τα πω στα δανέζικα, θα τα πω στα ολλανδικά και θα σας πω και αυτά που θα έλεγα κι εγώ. Ε, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Κόχ, πολύ καλή έκθεσή του. Γι' αυτό 7 ε, τροπολογίες έχω κάνει με τη διπλή μου ιδιότητα, γιατί είμαι και σκιώδη ηγητή στην ΙΜΚΟ, ο συνάδελφος Ρόντε 18 τροπολογίες. Αυτό <laughs> δείχνει ε, το κατά πόσο είμαστε ικανοποιημένοι, πόσο μπορεί να βελτιωθεί η έκθεση. Και κάθε θύμα τροχαίου είναι ένα θύμα που δεν πρέπει να υπάρχει. Στη χώρα μου, Δυστυχώ, από το 2014 και μετά έχουν αυξηθεί οι νεκροί στην άσφαλτο και πραγματικά πρέπει να λάβουμε μέτρα σαν αυτά που συζητάμε σήμερα εδώ. Ε, η πρώτη ενότητα τροπολογιών μου ε, βάζει πραγματικά την εστίαση στην Ευρώπη ε, των φιλοδοξιών. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ηγέτης παγκοσμίως στην αδική ασφάλεια. Με υψηλότερες προδιαγραφές έτσι τελικά θα έχουμε λιγότερα θύματα από τροχέα. Θα πρέπει αυτό να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς γραφειοκρατία, με ε, τη σωστή προσέγγιση από τα διδάγματα του παρελθόντος και από τις βέλτιστες πρακτικές όλων μας στα διάφορα κράτη-μέλη. Περί τίνος πρόκειται εδώ, εναρμόνιση ακούμε των μέτρων και μια δικιά μου τροπολογία έχει να κάνει με αυτό. Το είπε και η κυρία Σενάλοβα για τη συγκεντρώση ενοπνεύματο στο αίμα που επιτρέπονται. Πραγματικά χρειάζεται εναρμόνιση, αλλά ε, να φροντίσουμε οι αυστηρότερες ρυθμίσεις που αποδίδουν στην Ευρώπη να δώσουν το καλό παράδειγμα και στα άλλα κράτη και όχι να χαλαρώσουμε ε, ε, από τις αυστηρότερες ρυθμίσεις μας. προσωπικά έχω να προσθέσω το εξής πιστεύω ότι το ενόπνευμα δεν συμβαδίζει και δεν παντρεύεται με το τιμόνι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα πρέπει λοιπόν να τίνουμε προς το μηδέν ε, στη συγκέντρωση ενοπνεύματος στο αίμα. Και ας πούμε ιδιαίτερα για την τοπική κυκλοφορία ε, σε παραμεθόριες περιοχές είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει στους πολίτες ότι έχουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για να μειωθεί ο αριθμός των θυμάτων αλλά ε, ό,τι αφορά τη συγκέντρωση του αλκοόλα, τι να κάνουμε, έχουμε διαφορές στην εθνική νομοθεσία και δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε ενιαία. Ένα άλλο θέμα, το είπα και στην ΕΜΚΟ για άλλη τροπολογία, αρνητικό παράδειγμα, μας κάνει εντύπωση ότι λέει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ένα στα πέντε αυτοκίνητα είναι λιγότερο ασφαλές από ό,τι λένε οι μελέτες και δοκιμές. Ένα στα πέντε. Και οι καταναλωτές συχνά παραπληροφορούνται. Γιατί δεν τους ενημερώνουν για την πραγματική ασφάλεια που παρέχει το ε, αυτοκίνητο. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα τεστ που λέγεται Euro NCAP και δίνει ε, αστέρια αλλά πάντα δεν συμβαδίζουν αυτά και υπάρχουν και ε, κάποιες ε, αιτιάσεις ε, για απάτες τύπου Dieselgate. Όταν ένας καταναλωτής αγοράζει ένα αυτοκίνητο που θέλει να είναι ασφαλές, κοιτάει πόσα αστέρια εμφανίζει στις δοκιμές Και αυτό αφορά διάφορε χώρε και τη δική σα ε, πρόεδρα και την Αυστρία, τη Γερμανία κτλ. Συμφωνώ με τις διάφορες τροπολογίες συναδέλφων 124-125 που έχω βάλει και εγώ με άλλους συναδέλφους ε, ε, σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και θα πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση της δυνατότητας ε, παροχής μαθημάτων από κάποιες σχολές οδηγών και κάποιους δασκάλους. Υπάρχουν διάφορα συστήματα που αναφέρουν τις τροπολογίες 145 μέχρι 169 για τα ευφύ συστήματα πέδησης ή οδήγησης θα πρέπει να δούμε ε, ποια είναι η αποτελεσματικότητα. Εξ ονόματος του δικού μας ε, φιλελεύθερου ε, εισηγητή, συντάκτη μάλλον σκιώδη, του κυρίου Ρόντε, πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το σχέδιο και έστω και ένα θύμα είναι ένα θύμα που δεν θα πρέπει να υπάρχει. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κράμερ παρακαλώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας και την ομάδα του για την καλή συνεργασία. Ε, υπόθηκαν ε, ήδη αυτά που θέλω να πω. Έχουν υιοθετηθεί πολλές τροπολογίες ε, στις συμβαστικές και δικές μας των Πρασίνων και σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, που λαμβάνετε υπόψη και τους πιο ασθενείς χρήστες, τους πιο αδύναμους χρήστες μάλλον των δρόμων μας που είναι οι πεζοί και οι ποδηλάτες. Ε, και από εκεί είναι τα περισσότερα θύματα και ξέρουμε ότι αυξάνεται ο ρυθμός των θυμάτων. Παρόλο που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε για οδική ασφάλεια, ε, να μην εστιάζουμε μόνο στα αυτοκίνητα. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα και λύσεις υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται και να είναι δεσμευτικές. Τώρα μια απλή ενθάρρυνση προφανώς είναι μια τρύπα στο νερό. Υπάρχουν κάποια σημεία που χωράνε βελτίωση θα πρέπει να καταλάβουμε πώς μπορούν να απενεργοποιούνται και αν μπορούν να επενεργοποιούνται αυτά τα συστήματα. Αυτό να επιτρέπεται μένα, αλλά να είναι εξαίρεση. Δεν είναι δυνατόν να έχω ένα σύστημα βοήθησης και μετά να το κλείνω ε, για να τρέχω. Πιάσαν ένα στο Βερολίνο που πήγαινε με 150 χιλιόμετρα σε μια περιοχή που ήταν 30 χιλιόμετρα το όριο. Άμα έχει τέτοιο σύστημα και δεν μπορείς να το απενεργοποιήσεις, δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Ε, επίσης, συμφωνούμε ότι τα συστήματα δεν θα πρέπει να είναι απλούστατα ε, κάτι που θα μπορεί κανείς να αγνοεί ή να παραγνωρίζει. Η ασφάλεια θα πρέπει να είναι ε, ο κανόνας και οι εξαιρέσεις να επιτρέπονται μένα όταν είναι απολύτως απαραίτητα. Και τώρα απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να ακούσει, παρακαλώ, καλά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πότε θα έρθει επιτέλου καμιά νομοθετική πρόταση, γιατί αδρανεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό κάναμε εμεί την ε, έκθεση πρωτοβουλία. Αν είχατε φέρει πριν από δύο χρόνια πρόταση νομοθετική, δεν θα γινόταν η λεφτή συζήτηση και θα ε, αντιδρούσαμε στις δικές σας απαντήσεις. Αλλά επειδή χρόνο είναι χρήμα και δεν ε, μπορούμε να έχουμε και άλλες χρονοτριβές και είπαμε ότι κάθε νεκρός από τροχαίο είναι ένας νεκρός που δεν θα έπρεπε να χάνει τη ζωή του ε, με τάση αυξάνουσα παρόλο που εμείς συζητάμε ότι πρέπει να μειωθεί. Ένα θεώρηση που υποτίθεται ότι θα έρθει, υποτίθεται ότι θα έρθει, για να δούμε τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία και συνεχίζεται η συνεργασία. Ευχαριστώ κύριος Ερτούγκ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή. Πολλά σημαντικά, λέει ο κύριος Κόχ, και όποιος τον ξέρει τον συνάδελφο Κόχ, ε, ξέρει ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια παρακολουθεί αυτά τα θέματα και μας προειδοποιεί και δικαίως. Κοιτάξτε, θα πρέπει να τονίσουμε πάρα πολύ τα σημαντικότερα σημεία ε, για την οδική ασφάλεια. Δεν θα ήταν λάθος να πει κανείς ότι θα πρέπει να ξαναδούμε ε, τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στους αυτοκινητοδρόμους, των επαγγελματιών οδηγών και κυρίως η τήρηση των κοινωνικών διατάξεων και των εργατικών διατάξεων ε, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Εγώ δεν γνωρίζω τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα στα οποία αναφέρθηκε ο εισηγητής. Εγώ θα ισχυριζόμουν ότι ε, θα ήταν υπερβολική η κόπωση των οδηγών φορτηγών, αλλιώ ο άλλος δεν πάει επίτηδες να πέσει πάνω σε σταματημένα αυτοκίνητα σε μποτιλιάρισμα χωρίς να φρενάρει. Επίσης θεωρώ ότι η κατάσταση των υποδομών ε, συνεισφέρει πάρα πολύ στην ασφάλεια. Χρειάζεται συντήρηση ε, και των αυτοκινητοδρόμων και στις γέφυρες και σε άλλα σημεία της υποδομής, γιατί ακριβώς οι υποδομές συνεισφέρουν και στην ασφάλεια ή στη μη ασφάλεια ε, μιας διαδρομής. Όλοι γνωρίζουμε τη στιγμή που Έχουμε διάφορες πινακίδες που δεν καταλαβαίνεις πού σε στέλνουν. Σήμερα είναι πιο διάκριτες οι γραμμές στην ασφαλτό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα νέα συστήματα που σε, που εμποδίζουν να φύγεις από τη λωρίδα σου, έχουν πολύ μεγάλη σημασία να ανανεώνεται η δρόμη για να μπορεί να διαβάζει το χρώμα της λωρίδας, το μηχάνημα. Και όλα αυτά τα θύματα που θρυνούμε ή τα περισσότερα είναι στις πόλεις. Και αν δούμε ποιοι άνθρωποι είναι αυτοί που χάνουν τη ζωή τους, είναι οι πιο ευάλωτοι. Πεζοί, ποδηλάτες, άνδρες και γυναίκες γι' αυτό στο μέλλον θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη μέρημνα και σε εθνικό επίπεδο να κατασκευάζονται και να συντηρούνται πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, όλο και περισσότερο και μάλιστα να έχουν και περισσότερο χώρο και μεγαλύτερη θέση στην οδική κυκλοφορία οι ποδηλάτες και οι πεζοί. Το έχετε ξαναδεί αυτό σε κάτι πεζοδρομιάκια να προσπαθούν οι πεζοί να κυκλοφορούν και να καταβροχθίζουν τα αυτοκίνητα ε, όλο το χώρο. Και ο καθένα από εμά είναι ταυτόχρονα και πεζό και ποδηλάτη ή και πεζό και ε, οδηγό ιοταχή. Ε, και πολλά δυστυχήματα με ποδηλάτε και πεζούς ακριβώς οφείλονται σε συγκρούσεις των πιο ισχυρών. Δηλαδή όταν τρακάρει ένα φορτηγό με ένα γιοταχή την πληρώνει ο πλησιέστερος ποδηλάτης ή πεζός. Θα πρέπει να επενέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ομοθεσία. Ας πούμε, στα φορτηγά θα πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένη η θάλαμη οδήγηση καμπίνες με καλύτερη ορατότητα. Γιατί υπάρχει η περίφημη αυτή τυφλή γωνία στα φορτηγά που δεν βλέπουν πραγματικά τους ποδηλάτες ή τους ε, πεζούς ε, από την καμπίνα οι οδηγοί. Και στα ΙΟΤΑΧΗ επίσης θα πρέπει να είναι έτσι οι προφυλακτήρες, ώστε ακόμα και αν ε, συγκρουστείς με ποδηλάτη ή αν χτυπήσει ένα πεζό, να μην ε, είναι αυτόματα θύμα ε, του τροχαίου. Αν αναπατώμε μέχρι το 2020, θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να περιοριστούν σε 15.000 οι νεκροί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε νεκρός είναι νεκρός που δεν θα έπρεπε να είχε χάσει τη ζωή του, το επαναλαμβάνω και εγώ, θα πρέπει να φτάσουμε με τη βοήθεια όλων σε αυτούς τους στόχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Έρτουγκ. Στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Πίτερ Μπρότιες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Κόχ για την έκθεσή του και φυσικά σας ευχαριστώ για τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Πιστεύουμε ότι όλες πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Επομένως, θα είμαι σύντομος προς το παρόν. Δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις συμβαστικές τροπολογίες και τη συνεισφορά της Επιτροπής Ίμκο. Ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω, γιατί έχει να κάνει με ερώτηση που μας απευθύνθηκε για το πόσο φιλόδοξο είναι το χρονοδιάγραμμά μας και απαντώ λέγοντας ότι είναι κάτι που προσπαθούμε σκληρά, το δουλεύουμε εδώ και κάποιο καιρό χρειαζόμαστε τη συνεισφορά μεγάλου αριθμού εμπλεκόμενων φορέων από τα δικαιώματα των πολιτών, από το, τον χώρο της ασφάλειας στις μεταφορές, αλλά και από τη βιομηχανία και τον κλάδο εν γέννη. Δεν εξετάζουμε ένα-δυο μέτρα μεμονωμένα, εξετάζουμε μια μεγάλη δέσμη μέτρων ε, αλλάζει βέβαια αναλόγως με το πώς το μετράει κανείς, αλλά ε, άνετα και εύκολα είναι ασφαλής ο ισχυρισμός να πούμε ότι τουλάχιστον 20 μέτρα εξετάζονται και άπαξ και τα υιοθετήσουμε ή τα προτείνουμε, θα είμαστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχουμε ένα τόσο φιλόδοξο πακέτο, μια τόσο φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την προστασία του ατόμου. Και ε, οριστικοποιούμε την μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων πολύ στενές προθεσμίες. Θέλουμε να έχουμε πρόταση έτοιμη μέχρι το πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσετε να με συνοδεύσετε σε αυτή την αναμονή ε, και να σας διαβεβαιώσω ότι θα αξίζει το κόπο. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, μας ξαναλέτε τις ημερομηνίες Άκουσα το πρώτο εξάμεινο του 2018 ή το δεύτερο εξάμεινο για πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακόμα καλύτερα, το πρώτο τρίμηνο, κυρία Πρόεδρε, το πρώτο τρίμηνο του 2018. Πολύ ωραία. Όλοι είναι μάρτυρες λοιπόν, σας άκουσαν. Αυτοί οι μάρτυρες. Πρέπει να πάρουμε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2018. Το σημειώνουμε και θα το παρακολουθούμε εκ του συνέγγυς. Ο κύριος Κόχο, εισηγητής, έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και πάλι για τις προτάσεις και τις ε, υπόλοιπες συζητήσεις. Παρ' όλα αυτά όμως να κοιτάξουμε το θέμα. Διάσωση ζώων λέει. Ε, μεγαλύτερη ασφάλεια των αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Τα αυτοκίνητα μας ενδιαφέρουν. Εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω είναι πολύ ωραία και καλά και με χαρά να τα βάλω, αλλά δεν μπορώ. Θα υπάρξουν και άλλες εκθέσεις πρωτοβουλίες για τα άλλα θέματα που δεν έχουν άμεση ασφάλεια, με, ε, σχέση μάλλον με την ασφάλεια των αυτοκινήτων. Αυτό μπορεί να το αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο κύριος Λοτόφσκι μίλησε για τους παραγωγούς, γιατί δεν θα πρέπει μόνο οι κατασκευαστές ε, και οι ασφάλειες να συμμετέχουν, αλλά και οι αυτοκινητοβιομηχανίες. εμείς θα ορίσουμε όμως ε, αν θα είναι υποχρεωτικό όχι. Ο κύριος Πανμέλη για έγκαιρη ε, ενημέρωση και το Euro NCAP, ναι δεν το είχα συμπεριλάβει γιατί όχι να βάλουμε και αυτή την παράμετρο. Ο κύριος Κράμερ ζήτησε και πάλι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να φέρει την νομοθεσία για τον κανονισμό για τη γενική ασφάλεια. Απαντάει λίγο τα όσα ζητήσατε, περίμενα και εγώ την απάντηση αυτή. Αγαπητέ Ισμαήλ Ερτούκ, δεν ξέρω, θα πρέπει στη συγκεκριμένη έκθεση να συζητήσουμε για συνθήκες εργασίας και τήρησή τους. Πρόκειται για την ασφάλεια των αυτοκινήτων. Δεν αφισβητώ αυτά που λέτε, αλλά εδώ θα πρέπει να το βάλουμε, να τον δούμε ε, στη συνεδρίαση των σκεδών εισηγητών. προστασία, προφυλακτήρες για προστασία από τη σύγκρουση, παθητική ασφάλεια κτλ. Έτσι ώστε να προστατεύονται και οι πιο ευάλωτοι όπως είναι οι ποδηλάτες και οι πεζοί. Όταν πραγματικά απέλθει η σύγκρουση, ε, αν δεν μπορεί αυτή να αποφευχθεί με τα διάφορα συστήματα, ε, καλώς να είναι έτσι προφυλακτήρες ώστε να μην τραυματίζουν χειρότερα. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ενεργητική ασφάλεια και όχι η πασιτική υποθετική, να μην γίνει το τρακάρισμα, όχι το τι θα συμβεί μετά. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup, monsieur. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κόχα. Στις 12 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε στις 9 η ώρα το πρωί. Και σε θυμίζω επίσης ότι στις 11 Οκτωβρίου στις 10 η ώρα το πρωί στα πλαίσια της Επιτροπής μας θα λάβει χώρα μια δημόσια ακρόαση του κυρίου Ζοντόντα, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη, αρμόδιος για την οδική ασφάλεια και ο οποίος θα μπορέσει με τη σειρά του να μας πει ποιε είναι οι βέλτιστε πρακτικέ σε διεθνέ επίπεδο και ποιε από αυτέ θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σα ευχαριστώ πολύ. Α περάσουμε στο επόμενο σημείο τώρα τη ημερήσια διάταξη, Παρουσίαση από τη Γενική Διεύθυνση κινητικότητα και Μεταφορών της πρότασης για την αθεώρηση του κανονισμού 868 του 2004 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις ενέργειες μεταφορές. Καλό τώρα τον κύριο Φιλίπ Κορνελής. Α, είστε ήδη εδώ. Καλησπέρα σας κύριε Φιλίπ Κορνελής. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Θα σας δώσω το λόγο για 10 λεπτά και στη συνέχεια θα ακούσουμε και τον εισηγητή μας, τον κύριο Πίπερ. Έχετε το λόγο και για άλλη μια φορά καλωσορίστε στην Επιτροπή μας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Έχω παρουσιάσει μια σειρά διαφανειών προκειμένου να σα παρουσιάσω την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Καταρχά, σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μα δώσετε τη δυνατότητα να κάνουμε τη σημερινή παρουσίαση. Καταρχάς, προτού περάσουμε στι λεπτομέρειες τη σχετική πρόταση, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη αυτή πρόταση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής μας για τις αεροπορικές μεταφορές, η οποία υιοθετεί την εξή οπτική γωνία, ότι οι αεροπορικέ μεταφορέ είναι πάρα πολύ σημαντικέ όχι μόνο ω κλάδο, αλλά και ω φορέα παροχή υπηρεσιών και στου υπόλοιπου οικονομικού κλάδου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η βασική ιδέα τη στρατηγική εκείνη που εγκρίναμε το Δεκέμβριο του 2015, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η αεροπορία θα συνεχίσει να πληρεί το ρόλο της στα πλαίσια της νέας οικονομίας και ότι θα μπορεί τελικά να κερδίζει και νέες αγορές αλλά και να τονώνει περισσότερο τις τοπικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα ερωτήματα που μας έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δούμε πώς θα καταφέρουμε να διατηρήσουμε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο για τη δική μας την αεροπορία, η οποία θα πρέπει να συνδέεται με τις υπόλοιπες αεροπορικές μεταφορές που λαμβάνουν χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι έχουμε πολλούς κανονισμούς αυτή τη στιγμή και διάφορες πρωτοβουλίες στον τομέα της αεροπορίας. Θα έλεγα πάντως ότι μια πιο πρόσφατη πρωτοβουλία είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια ανοιχτή και συνδεδεμένη Ευρώπη από πλευράς αεροπορικών μεταφορών. Την ανακοίνωση αυτή την εγκρίναμε τον Ιούνιο του 2017. Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας αυτής προβλέπεται μία σειρά υποπρωτοβουλειών, αν μου το επιτρέπετε, δηλαδή κατευθύριες γραμμές όσον αφορά τον έλεγχο, Επίσης, κατευθυντήρες γραμμές όσον αφορά τις υποχρεώσεις των δημοσίων φορέων για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών, προκειμένου να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε την όλο και αυξανόμενη κίνηση στους ευρωπαϊκούς ουρανούς. Επίσης, βελτιώσεις και βιωσιμότητα όσον αφορά τη διαχείριση νέας κυκλοφορίας, ATM, και έπειτα υπάρχει και αυτός ο γενικότερος στόχος της βελτίωσης και της ενίσχυσης της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διεθνή φόρα αεροπορίας. Και στα πλαίσια λοιπόν της πρωτοβουλίας αυτής έχουμε και τη συγκεκριμένη σημερινή πρόταση για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Από αυτού θα επικεντρωθούμε σήμερα και ελπίζω ότι ε, μπορείτε και εσείς εν συνεχεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αρχίσετε να εξετάζετε την ε, πρόταση αυτή. Ποιο είναι το γενικότερο υπόβαθρο τώρα για την πρόταση αυτή που έχει να κάνει με την ανταγωνιστικότητα των αεροπορικών μεταφορών. Λοιπόν, ας δούμε καταρχάς το εξής. Υπάρχει μία σύνδεση ανάμεσα στην ε, συνδεκτικότητα συνδεσιμότητα μάλλον με συγχωρείτε, συνδεσιμότητα των αεροπορικών μεταφορών. Υπάρχει άμεση λοιπόν σύνδεση τη συνδεσιμότητα αυτή και τη οικονομική ανάπτυξη. Έχουμε δει για παράδειγμα ότι ένα 10% αύξηση στην συνδεσιμότητα αεροπορικών μεταφορών σε μια περιοχή οδηγεί σε περισσότερο εμπόριο, αύξηση κατά 4% όσον αφορά τα βασικά κεντρικά γραφεία των μεγάλων επιχειρήσεων και οδηγεί επίσης σε πολύ σημαντική αύξηση του ΑΕΠ. Και όντω η συνδεσιμότητα την τελευταία περίοδο έχει αυξηθεί πάρα πολύ σημαντικά και έχουμε 23.000 πλέον πτήσει σε καθημερινή βάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ήταν μόνο 10.000 οι πτήσει όταν δημιουργήθηκε, όταν ολοκληρώθηκε η εσωτερική αγορά πριν από 25 χρόνια δηλαδή. Βλέπετε εδώ πέρα μία σειρά γραφικών παραστάσεων. Στόχος μας εδώ πέρα είναι να καταφέρουμε να σας δείξουμε καλύτερα τις πολλές διαφορετικές μορφές που μπορεί να πάρει η περίφημη αυτή συνδεσιμότητα. Έχουμε άμεση συνδεσιμότητα μεταξύ πόλων. Για παράδειγμα, βλέπετε εδώ πέρα στους χάρτες που έχετε ενώπιόν σας, πάνω αριστερά για παράδειγμα, βλέπετε τις δυνατότητες συνδεσιμότητας από τη Λισαβόνα με πράσινο. Έχουμε τους αερομεταφορείς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κόκκινο έχουμε τη στεσιμότητα που παρέχουν μη ευρωπαϊκοί φορείς, ενώ με μπλε έχουμε του αερομεταφορείς εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά λάθος έκανα. Άμα συγχωρείτε, με μπλε χρώμα βλέπουμε τι ευρωπαϊκέ αεροπορικέ εταιρείε και πράσινο του αερομεταφορείς εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, η Πορτογαλία έχει πολύ καλή σύνδεση με τη Βραζιλία. Δεν μα προκαλεί εντύπωση αυτό. Ένα άλλο παράδειγμα που βλέπετε εδώ είναι πάνω δεξιά. Θα σα δώσουμε προφανώ τι διαφάνειε αυτές, γιατί μάλλον δεν είναι τόσο ευανάγνωστε. Βλέπετε εδώ πέρα τις δυνατότητες συνδεσιμότητας μέσω αεροπορικών μεταφορών από το Ταλίν. Από το Ταλίν προς την Ιαπωνία, για παράδειγμα. Εδώ βλέπουμε πάρα πολύ καλά περιπτώσεις έμεσης συνδεσιμότητας. Για άλλη μια φορά βλέπετε εδώ πέρα με τα διάφορα χρώματα ότι η έμεση συνδεσιμότητα είναι πολύ σημαντική και ουσιαστικά είναι ο μόνος τρόπος για να πάει κανείς από την Εστονία στην Ιαπωνία. Παράλληλα υπάρχουν όμως και πολλές συναλλακτικέ οι οποίες παρέχονται τόσο από αερομεταφορείς εντός Ένωσης όσο και αερομεταφορείς εκτός Ένωσης. Στόχος μας είναι να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερες εναλλακτικέ και όσο δυνατόν μεγαλύτερο επίπεδο ανταγωνισμού όσον αφορά τις διασυνδέσεις αυτές, γιατί όπως σας είπα λειτουργούν προς το συμφέρον τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων εν προκειμένου για την Εστονία. Έχουμε κόμβους εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, στο κάτω μέρος διαφάνειας βλέπετε δύο τέτοια παραδείγματα. Βλέπετε τις δυνατότητε συνδεσιμότητας κάτω δεξιά που έχουμε από τον κόμβο του Παρισιού. Βλέπετε όλες τις πόλεις οι οποίες εξυπηρετούνται μέσω πτήσεων από το Παρίσι. Μπορεί λοιπόν κανείς ερχόμενος στο Παρίσι στη συνέχεια να μεταβεί σε όλους αυτούς τους προορισμούς. Στα αριστερά βλέπετε τις δυνατότητες άμεσης συνδεσιμότητας από τη Βαρσοβία. Και για άλλη μια φορά βλέπετε εδώ πέρα ότι υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης τόσο ευρωπαϊκών όσο και μη ευρωπαϊκών αερομεταφορέων. Για μας όλες αυτές οι μορφές έμεσης ή άμεσης δεσιμότητας είναι πολύ σημαντικές και πραγματικά θέλουμε να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες ανταγωνισμού τόσο εκτός όσο και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, πότε απειλείται αυτός ο ανταγωνισμός στα εσωτερικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξέρετε ότι έχουμε τα απαραίτητα μέσα και εργαλεία. Έχουμε την εσωτερική αγορά, έχουμε τους κανόνες ανταγωνισμού, έχουμε τους κανόνες πρόσβασης στην αγορά, δεν επιτρέπεται η διακριτική μεταχείριση μεταξύ αερομεταφορέων σε ένα συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Επομένως, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τα απαραίτητα μέσα για να βάλουμε κατά αυτή τη διακριτική μεταχείρισης. Εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση όμω τι κάνουμε. Ενδεχομένω τα πράγματα να μην είναι τόσο εύκολα σε περίπτωση Διακριτική μεταχείρισης ή πρακτικών που εισάγουν διακρίσει. Έχουμε και περιπτώσεις αθέμητων πρακτικών, έχουμε και περιπτώσεις πρακτικών που εισάγουν διακρίσει οι οποίε προέρχονται από χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία μείωση του ανταγωνισμού στι συγκεκριμένε αυτέ τρίτε αγορέ. Και μακροπρόθεσμα θα μπορούσαν ακόμα και να μειώσουν τον αριθμό των αερομεταφορέων που μπορούν να δραστηριοποιούνται σε αυτέ τι αγορέ και άρα αυτό με τη σειρά του μειώνει και τη συνδεσιμότητα. Και όταν είναι χαμηλότερο ο ανταγωνισμό, είναι μικρότερε και λιγότερε επιλογέ και αυξάνονται όπω ξέρετε οι τιμέ και οι ναύλοι. Επομένω αυτό είναι ιδιαίτερα αρνητικό και για τους εμπλεκόμενους αερομεταφορείς, αλλά και γενικότερα για τους Ευρωπαίους πολίτες και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα, στον τομέα της αεροπορίας, σε αντίθεση με άλλους τομείς, δυστυχώς δεν υπάρχουν δυνατότητες αναδίπλωσης σε διεθνείς κανόνες. Δεν προβλέπει τίποτα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου για την διεθνή αεροπορία. Έχουμε τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτική Αεροπορία, ο οποίο όμω και πάλι δεν διαθέτει ξεκάθαρου κανόνε όσον αφορά το ζήτημα του ανταγωνισμού. Συνεπώ, δεν υπάρχει ένα παγκόσμιο καθεστώ προστασία του ανταγωνισμού. Επίση, βλέπουμε ότι περισσότερε διμερεί συμφωνίε αεροπορία δεν καλύπτουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με αθέμητο ανταγωνισμό, αθέμητε πρακτικέ ή ακόμα και αν το κάνουν, το κάνουν με τόσο ήπιο τρόπο που τελικά δεν μπορούμε εμεί να εφαρμόσουμε στην πράξη κανένα κανόνα. Και αυτό το λόγο θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμπληρώσουμε την εργαλειοθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα του εμπορίου με μέσα εκείνα τα οποία μπορούν να προασπίσουν το εμπόριο, τον ανταγωνισμό και ότι θα πρέπει να μπορούμε και εμείς να επεμβαίνουμε όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Έχουμε βασίσει την πρότασή μας αυτή, την όλη τη λογιστική μας, σε παραδείγματα που έχουμε σε άλλους τομείς και ιδίω στα πλαίσια του κανονισμού για τα εμπόδια στο εμπόριο. Συνεργαστήκαμε δηλαδή εκεί πέρα με συναδέλφους από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου για να δούμε τι έχουν κάνει αυτοί για να προστατεύσουν το εμπόριο και τις υπηρεσίες σε άλλους τομείς, εκτός αεροπορίας βέβαια. Θελήσαμε ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε τις βασικές έννοιες που έχουμε στο εμπόριο και τις βασικές διαδικασίες που ήδη έχουμε στο εμπόριο, προκειμένου να δούμε αν μπορούμε να εφαρμόσουμε τις ίδιες πρακτικές και στην αεροπορία. Συνεργαστήκαμε λοιπόν με τους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και Ανταγωνισμού για την εκπόνηση αυτής της πρότασης. Αυτή η πρόταση κανονισμού, μελλοντικού κανονισμού ελπίζω, θα είναι μέρος της γενικότερη εργαλειοθήκης που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλουμε να έχουμε και πιο παγκόσμιε, αν θέλετε λύσει, λύσει οι οποίε να μπορούν να λειτουργήσουν και σε διεθνέ επίπεδο. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν στα πλαίσια του ΙΚΑΟ να ενισχύσουμε του ήδη εγκεκριμένου εκεί κανόνε. Θεωρούμε ότι με την πρόταση αυτή μπορούμε να συμπληρώσουμε τι διμερεί μα συμφωνίε, είτε είναι ευρωπαϊκέ συμφωνίε, είτε είναι συμφωνίε μονομένων κρατών μέλων τη Ένωση. Και βέβαια ο κανονισμό αυτό δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει τι φυσιολογικέ συνθήκε συνταγωνισμού στην αγορά. Ουσιαστικά οι αερομεταφορεί θα εξακολουθούν να είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την ανταγωνιστικότητά τους οφείλουν να παρέχουν καλά προϊόντα και υπηρεσίες σε θεμητές τιμές. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν θέλουμε να επέμβουμε στα πεδία του ανταγωνισμού. Σε καμία περίπτωση λοιπόν ο κανονισμός αυτός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προστατευτικούς ε, σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να δώσει πλεονεκτήματα σε κάποιους αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανταυτού ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει αποτρεπτικό μέσο όπως και τα περισσότερα μέσα προστασίας του εμπορίου. Ξέρετε ότι τα μέσα αυτά σπάνια χρησιμοποιούνται, μόνο και μόνο το ότι υπάρχουν όμως πολύ συχνά οδηγεί στο να αποτρέπονται ορισμένοι από το να χρησιμοποιήσουν τέτοιες αθέμητες πρακτικές. Ξέρετε ότι πολύ συχνά, ακόμα και όταν εμφανίζονται κάποιε υποψίε τέτοιων αθέμητων πρακτικών κινητοποιούνται αυτόματα αυτά τα μέσα προστασία του εμπορίου και του ανταγωνισμού. Άρα είναι καλό να υπάρχουν έστω και αποτρεπτικά. Τώρα, να σας δώσω κάποιες λεπτομέρειε όσον αφορά την πρόταση αυτή καθεαυτή. Τι προσπαθούμε να καλύψουμε. Καταρχά, στις περιπτώσεις εκείνες όπου έχουμε μία παραβίαση διεθνών υποχρεώσεων σε τρίτη χώρα, υποχρεώσεων που έχει δηλαδή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή αν έχουμε πρακτικές που έχουν επιπτώσει στον ανταγωνισμό, δηλαδή πρακτικέ που εισάγουν διακριτική μεταχείριση προσπαθούμε να καλύψουμε τις περιπτώσεις εκείνες όπου έχουμε αερομεταφορείς Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και άλλους αερομεταφορείς και μόνο στην περίπτωση εκείνη βέβαια που οι πρακτικές αυτές, οι παραβιάσεις αυτές απειλούν ή προκαλούν πραγματικά ζημία σε αερομεταφορείς. Έχουμε λοιπόν δύο βασικές περιπτώσεις όπου μπορούμε να λάβουμε δράση. Όταν αφαιτούνται διεθνείς υποχρεώσεις ή όταν ακολουθούνται πρακτικές ε, που εισάγουν διακρίσεις και βάλουν κατά του θεμητού ανταγωνισμού. Πώς λειτουργεί τώρα το σύστημα αυτό στην πράξη. Στην πρότασή μας λέγεται ότι οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν από διάφορους φορείς, καταρχάς από τέτοια τα κράτη-μέλη, από αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ενώσεις αερομεταφορέων της Ένωσης ή αυτεπάγγελτα μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με δική της πρωτοβουλία να υποβάλει μια καταγγελία όταν δει ότι άλλοι φορεί στην αγορά διστάζουν να υποβάλουν μια καταγγελία. Στη συνέχεια, η καταγγελία αυτή θα πρέπει να φτάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απαραίτητη αιτιολόγηση. Δεν αρκεί δηλαδή να μας στείλετε απλώς μια πρόταση που θα λέει «Κοιτάξτε την περίπτωση αυτή». Περιμένουμε έναν πλήρη φάκελο που θα έχουμε αν μη τι άλλο κάποια πρώτα αποδεικτικά στοιχεία δεν, δεν μπορούμε να βασιστούμε σε, με τίποτα σε φήμες ή απλώς σε κάποια άρθρα του τύπου. Πρέπει να δούμε αν πραγματικά υπάρχει βάση προκειμένου να κινηθεί έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πρέπει βέβαια να δούμε αν η έρευνα αυτή όντως συνάδει με το γενικότερο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινάει λοιπόν η διαδικασία της έρευνας εν συνεχεία. Στο κείμενο προτείνουμε ότι η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο ετών και αν λάβει λιγότερο χρόνο τόσο το καλύτερο. Θεωρήσαμε πάντως ότι θα πρέπει να υπάρχει μία συνολική προθεσμία προκειμένου να υπάρχει και απαραίτητη νομική ασφάλεια και προβλέπεται και μια διαδικασία επίγουσας ανάγκης όπου μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα. Προβλέπεται επίση ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη και εμπειρογνώμονε από τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στι έρευνε αυτέ. Ξέρετε ότι πολλέ φορέ υπάρχουν εμπειρογνώμονε σε κράτη-μέλη που γνωρίζουν πολύ καλά τι συγκεκριμένε αυτέ περιπτώσει και θα μπορούσαν να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια καλή έρευνα. Και Βέβαια υπάρχουν και πολύ σημαντικές ισχυρές ρήτρε στην πρόταση αυτή όσον αφορά το δικαίωμα υπεράσπισης και το δικαίωμα όλων των εμπλεκόμενων φορέων και από τι δύο, από τις δύο πλευρές να έχουν το δικαίωμα ακρόασης. Η εκτίμησή μας στο τέλος πρέπει σε κάθε περίπτωση να πραγματοποιείται με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά περιστατικά. Δηλαδή, θα καλέσουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να υποβάλουν αποδεκτικά στοιχεία, αλλά θα πρέπει εμείς να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα βάσει των όσων μας προτείνονται. Αν δεν, υπάρχουν, λοιπόν, αν δεν υπάρχει συνεργασία από κάποιους εμπλεκομένους, τότε αυτό θα είναι εις βάρος προφανώς, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ολοκληρώσει ούτως ή άλλως την έρευνά της βάσει των αποτυχητικών στοιχείων που έχουν υποβάλει οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορεί. Τώρα, τι είδου δράση μπορεί να αναλυφθεί. Όπω είπα πριν από λίγο, σε κάθε περίπτωση ευνοούμε μία διαπραγματευτική λύση, μία λύση που θα έχουμε διαπραγματευτεί με τα εμπλεκόμενα μέρη. Μπορεί να μην έχουμε συμφωνίε με όλε τι τρίτε χώρε, πάντω θα συνομιλήσουμε μαζί του πρώτα και θα προσπαθήσουμε μέσω τη συνεργασία να καταλήξουμε σε μία λύση. Και αυτό μπορεί να γίνει ακόμα και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έρευνας. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν όλες τις δυνατές λύσεις προτού καταλήξουμε τελικά σε συγκεκριμένα μέτρα ιδίως όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εκείνες συμφωνίες που ξέρω ότι προβλέπουν πολύπλοκες διαδικασίες όσον αφορά την επίλυση διαφορών. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα εξαντλήσουμε όλες αυτές τις νομικές δυνατότητες βάσει των συμφωνιών αυτών προτού καταλήξουμε σε κάποια επαναρθωτικά μέτρα. Όσον αφορά τώρα τις διμερείς συμφωνίες των κρατών μελών, όπου υπάρχει εκεί πέρα μια θέμητη ενδεχομένω πρακτική, προτού λάβουμε πάλι δράση στο τέλος της ε, έρευνας, θα πρέπει να απαντήσουμε θετικά σε τρία ερωτήματα. Πρώτον, υφίσταται όντως διακριτική μεταχείριση. Δεύτερον, υφίσταται όντως ζημία σε βάρος αερομεταφορέα της Ένωσης ή σε βάρος πολλών αερομεταφορέων της Ένωσης. Και τέλος, υπάρχει όντως αιτιώδη συνάφη ανάμεσα στην πρακτική αυτή που εισάγει διακρίσεις και την ζημία αν απαντήσουμε θετικά και στι τρει αυτέ ερωτήσει βάσει αποδεκτικών στοιχείων, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προτείνει πραγματικά μέτρα προκειμένου να επανορθώσει, να αντισταθμίσει τη ζημία που έχει λάβει η χώρα. Μέτρα αντισταθμιστικά. Σε καμία περίπτωση τα μέτρα αυτά δεν θα είναι τιμωρητικά. Στόχος μας θα είναι για παράδειγμα να επιβάλλουμε ένα χρηματικό πρόστιμο το οποίο θα αντιστοιχεί στη ζημία που έχει υποστεί που έχει υποστεί ένα αερομεταφορέα. Και κατά αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αντισταθμίζεται πάλι η κατάσταση, εξορροπεί την κατάσταση στην αγορά και προφανώ το μέτρο αυτό, αν προκειμένου το πρόστιμο, θα ανασταλεί όταν η διακριτική μεταχείριση πάυσει να ισχύει. Τα μέτρα αυτά δεν θα εφαρμόζονται αυτόματα, με το τέλος δηλαδή της έρευνας, ακόμα και αν απαντήσουμε θετικά στο τέλος της έρευνας τα τρία αυτά ερωτήματα, δεν πρόκειται αυτόματα να αρχίσουν να ισχύουν τα επανορθωτικά μέτρα, πάλι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεδριάσει και να δει τελικά αν η ανάληψη δράση δεν είναι τελικά πιο επιζήμια από το να μην αναλυφθεί δράση, από το να μην επιβληθούν μέτρα. Ξέρετε ότι μερικές φορές έχουμε δει και από άλλους οικονομικούς τομείς ότι το συμφέρον των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, των καταναλωτών ενδεχομένως να είναι υψηλότερο τελικά από τη ζημία που μπορεί να έχει υποστεί ένας αερομεταφορέας. Στην περίπτωση αυτή, όπως έχουμε δει και στα πλαίσια του κανονισμού για τα εμπόδια στο εμπόριο, μπορεί να μην αναλάβουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή δράση, γιατί θεωρούμε ότι προέχει το συμφέρον των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και στην περίπτωση που θα αναλάβουμε δράση, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θέσουμε αυτού ή τα κράτη-μέλη σε μια τέτοια θέση που τελικά θα παραβιάζουμε τη συμφωνία που έχουμε υπογράψει με την συγκεκριμένη τρίτη χώρα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να συμβεί κάτι τέτοιο. Και βέβαια τα μέτρα αυτά θα πρέπει προφανώς να είναι αναλογικά και όπως σας είπα μπορούν μόνο να αντισταθμίσουν τη ζημία, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχουν κάποιον τιμωρητικό χαρακτήρα ή να ευνοούν τελικά ή να δίνουν πλεονέκτημα σε κάποιον αερομεταφορέα. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να έχουμε ίσες ευκαιρίες. Συνοψίζοντας λοιπόν, ο στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι έχουμε ανταγωνιστικές αγορές τόσο εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι έχουμε πρόσβαση στις αγορές χωρίς διακριτική μεταχείριση, όπως ακριβώς και οι αερομεταφορείς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να έχουν ε, συνθήκες χωρίς διακριτική μεταχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι πρέπει να γίνεται και με τις δικές μας τις ε, αεροπορικές εταιρείες. Θέλουμε βελτιωμένο ανταγωνισμό και συνδεσιμότητα και περισσότερες επιλογές για τους επιβάτες μας εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Merci. Ευχαριστώ. Κύριε Κορνέλης, μας ε, παρουσιάσατε ένα είδος οδικού χάρτη τρόπον την οδικού χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ξεκινήσει λοιπόν η συζήτηση τώρα. Ο κύριος Πίπερ, ο εισηγητής μας καταρχάς, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Κορνέλης. Πολύ σαφής ξεκάθαρη και πιστική παρουσίαση θα έλεγα ταυτόχρονα είναι γεγονός. Στις ενέργειες μεταφορές χωράει βελτίωση η υπόθεση του θεμητού ανταγωνισμού. Οι ρυθμίσεις που είχαμε για την αυθαίρετη τιμολόγηση σχεδόν ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. Ενώ σε άλλα κράτη της γης υπάρχουν αποτρεπτικά μέτρα, άλλα τα οποία δεν εφαρμόζονται μεν, ε, αλλά υπάρχουν. Βλέπε οι Ηνωμένε Πολιτείες και οι αερομεταφορείς προσέχουν όταν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία και τους απειλεί σε περίπτωση που κάνουν κάτι κακό. Πραγματικά λοιπόν εδώ χρειάζεται να δράσουμε. Πώς θα γίνει αυτό. Πρώτα με ήπιες διαδικασίες, το είπατε και εσείς ο ίδιος, διμερός, ε, συμφωνίες. Υπάρχει δυνατότητα επίλυσης διαφορών και διακανονισμού και νομίζω 90% για να μην πω 95% των προβλημάτων ε, μεταξύ κρατών ε, διεκπεραιώνονται με τον τρόπο αυτό. Υπάρχει στη συνέχεια ένα δεύτερο στάδιο όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ίδια εκείνη διαδικασία στον ΝΑΙΚΑΟ, μέσω δηλαδή παγκοσμίων συμφωνιών προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα που ανακύπτουν. Όλα αυτά τα πράγματα ήδη τρέχουν και λειτουργούν, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια εταιρεία στην Κίνα, τη Ρωσία, στον αραβικό χώρο ή κάπου που ε, προβαίνει σε διακρίσεις και περιορίζει κατά πολύ τα δικαιώματα προσγείωσης των ευρωπαϊκών εταιριών με, με άσχημες ε, χρονοθυρίδες, κακά ωράρια κτλ. Ή αν περιορίζονται δικαιώματα πτήσης με διάφορα καψόνια, γιατί υπάρχουν και τέτοια πράγματα και τα παρακολουθούμε ε, και τα παρατηρούμε. Αν αυτό γίνεται ο κανόνας, λέω λοιπόν, χρειαζόμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μέσο και ένα μέτρο αποτροπής. Αυτό προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Δεν πρόκειται ότι αυτό θα γίνει μεγάλη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό θα το συζητάμε ακόμα δεκαετίες. Πάντως είναι ένα αποτρεπτικό μέσο που υπάρχει και θέλω να καθησυχάσω λίγο τα αεροδρόμια που ανησυχούν, ε, μήπως περιορίσουμε τον ανταγωνισμό. Σε καμία περίπτωση. Είναι λίγες μεμονωμένες περιπτώσεις που θέλουμε να δείξουμε με κάποιες διαδικασίες ότι κοιτάξτε να δείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και κανόνες, έχει και μέσα, έχει και μέτρα και θα πρέπει να τα τηρούν οι αεροπορικές εταιρείε. Νομίζω θα το πετύχουμε στο μέλλον δεν σημαίνει ότι θα στραγγίξουν ή θα στεγνώσουν ολόκληρα αεροδρόμια ή ολόκληρες περιφέρειες, για να μην πω κράτη-μέλη, γιατί τα ακούμε και αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Το ξεκαθαρίζει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Λοιπόν, συμπέρασμα. Σε πρώτη φάση το βλέπω θετικά. Υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν προτείνει και κάποιοι συνάδελφοι και που χωράνε βελτίωση. Η δική μου πολιτική ομάδα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, θα κάνει κάποια πολιτική σίγουρα επισήμαση. Είμαι πολύ αισιόδοξο για τη συζήτηση και χαίρομαι. Αλλά να τονίσω ότι κατά την άποψή μου η συγκεκριμένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Που είναι η Πρόεδρος. Χάσαμε την Πρόεδρο. Κύριε Σγικέ, ευχαριστώ η κυρία Πρόης. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και σα, κύριε Κορνέλη, για την πολύ καλή αυτή πρόταση που μα παρουσιάσετε σήμερα με διαφάνεια. Και η δική μου πολιτική ομάδα, σοσιαλιστή και δημοκράτε, και στο παρελθόν μιλήσαμε για αφόρητες και απαράδεκτες καταστάσει ε, που επικρατούν στην εναέρια κυκλοφορία δεν έχουμε ένα σωστό θεμητό ανταγωνισμό, τακτικό ε, ανταγωνισμό, αλλά βλέπουμε διάφορες πρακτικές, διάφορες ε, τακτικές ε, του ποδαριού, διάφορες προσπάθειες εξαπάτησης. Αυτό είναι κάτι που αποδυναμώνει τις δικές μας εταιρείες στο διεθνή ανταγωνισμό και χαίρομαι πάρα πολύ που τώρα δημιουργούμε ένα μέσο ε, για να αμυνθούμε απέναντι σε στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού. Και ενθαρρύνω όλους τους ενδιαφερόμενους, αν δεν υπάρχει άλλος δρόμος, να καταφεύγουν σε αυτά τα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παγκόσμιος ε, οικονομικός πρωταγωνιστής και δεν μπορεί ε, κανένας να παραβιάζει τον ανταγωνισμό. Δεν συμφωνώ με κάποιους που λέγουν ε, ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε έγκριση μέτρων για να μην ε, έχουμε αντίπεινα. Οι επιχειρήσεις μας υφίστανται διακρίσεις με διάφορες ενισχύσεις που παίρνουν κάποιες άλλες εταιρείες. Θα πρέπει γρήγορα να έρθει ε, ο αντίστοιχο κανονισμός. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη ε, τα οποία κόπτονται κατά τα άλλα για τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την ελεύθερη αγορά, τα οποία καθυστερούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι μέτρα προστασίας απέναντι σε αθέμητο ανταγωνισμό δεν είναι τρόπος να εκδιώξεις από την αγορά ανεπιθύμητους ε, και μη δημοφιλείς ανταγωνιστές. Ε, θα πρέπει λοιπόν να μην έχουμε το αποτελέσματα που είναι αντίθετο από αυτό που επιδιώκουμε. Γιατί και ξένες εταιρείε είναι εταιρείε που έχουν εργαζομένου που λειτουργούν, που κυκλοφορούν και είναι εμπλουτισμό για τη δική μα αγορά στο βαθμό που λειτουργούν σωστά. Θα ήθελα λοιπόν να διαφυλαχθούν και τα ενδιαφέροντα και τα συμφέροντα των αερολιμένων και των ε, κατασκευαστών αεροσκαφών. Τις επόμενες ημέρες θα συναντηθούμε με τον κύριο Πίπερ, οι υπόλοιποι σκιώδεις ηγητές, για να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση από πλευρά της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος. Merci ευχαριστώ. Ο κύριος Στανίσκα έχει το λόγο. Τελίτσκα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Κορνέλης για την παρουσίαση αυτή. Θα ήθελα καταρχάς να υπογραμμίσω κάτι. Γιατί και οι λέξεις που χρησιμοποιούμε έχουν τη σημασία τους. Δεν είναι ένα εργαλείο προστασίας για μένα αυτό. Είναι ένα πρότυπο ταξιδιού που θεσπίδιζεται για να αντιμετωπιστεί η μία ανταγωνιστική ε, συμπεριφορά, μία συμπεριφορά η οποία δεν είναι φιλική προς τον ανταγωνισμό και η οποία δεν συνάδει και δεν είναι συμβατή ε, με τις πεπιθήσεις μας. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο ρόλος μας δεν είναι να εικάζουμε κατά πόσο υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, ούτε του τι ακριβώς σημαίνει αθέμητος ανταγωνισμός, γιατί υπάρχουν αρμόδιες αρχές να το αποφασίσουν αυτό. Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ρόλος μας σήμερα, από σήμερα και τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες είναι να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια νομοθεσία στα χέρια μας, η οποία να είναι η βέλτιστη δυνατή, θα δίνει τις καλύτερες δυνατές δικλίδες ασφαλείας θα δίνει ένα στέρεο εργαλείο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει να δράσει εάν το χρειαστεί. Ε, γίνομαι πλέον ασματικός, δηλαδή επαναλαμβάνομαι ξανά και ξανά, αλλά θέλησα πραγματικά να πάρω αυτό το χρόνο για να διευκρινίσω το ρόλο μας, γιατί έχει συμβεί στο παρελθόν σε λεπτά ζητήματα, σε ακαθόδη ζητήματα και κατανοώ ότι έχει υπάρξει και αθέμητος ανταγωνισμός αλλά ε, στο παρελθόν έχουμε εικάσει υπερβολικά πολύ και έχουμε πλειοδοτήσει του υπερβολικά πολύ στο ότι σίγουρα υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει ακολουθήσει πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις και νομίζω ότι έχει διαλέξει τη σωστή. Απεικονίζει η φυστάμενη νομοθεσία σε άλλους τομείς εκτός της αεροπλοείας και Ασχολείται δηλαδή με νομοθετήματα που έχουν αντέξει στη δοκιμή του χρόνου. Και ε, υπάρχουν ζητήματα που έχουν καταληφθεί με την νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις. Και αυτό είναι κάτι το θετικό. Επειδή η δουλειά μπροστά μας θα κρατήσει πολύ και θα είναι μακροχρόνια η εργασία μας. Θέλω να πω κάτι. Η αξιολόγηση επιπτώσεων δεν είναι πρώτης ποιότητας σε όλα τις τα θέματα και σε όλα τις τα στοιχεία ή τουλάχιστον δεν έχω πιστεί γι' αυτό ποιο αντίκτυπο θα έχει στη συνδεσιμότητα κάποιων περιφερειακών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό νομίζω ότι δεν έχει εξεταστεί με ισορροπημένο τρόπο στην έκθεση και στη μελέτη. Ίσως και αργότερα θελήσετε να τοποθετηθείτε για τη σχέση σας με το Συμβούλιο και πώς ε, διάκειται το Συμβούλιο εναντί της αξιολόγησης επιπτώσεων. Τούτων λεχθέντων δεν τα θεωρώ αυτά λόγο η δικαιολογία αφορμή για να ζητήσω από κάποιους από εσάς να ε, ε, έρθουμε σε αντιπαράθεση μαζί σας για το σχέδιο αυτό γνωμοδότηση, γιατί είναι καλό. Είναι απολύτως κατανοητός ο προληπτικός χαρακτήρας. Πολύ καλά καθορίσατε τα διάφορα ε, στάδια και φάσεις. Μέχρι δύο χρόνια και μέχρι, δύο, μέχρι ένα έτος σε επίγουσα κατάσταση είναι οι προθεσμίες και καλός. Όμως, οι δύο διαπραγματεύσεις για τις διμερείς συμφωνίες με κάποιους από τους ομολόγους μας προχωρούν και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό να το λάβει υπόψη της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ε, συμπεριλάβει αυτό που τη ζητήσαμε. Δηλαδή να δώσουμε προσοχή στις διμερείς σχέσεις και εδώ έχουμε και ένα άλλο εργαλείο αν η πρώτη επιλογή δεν δουλέψει γνωρίζουμε τι προτείνεται και τι γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης, αλλά δεν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε με λεπτομέρεια αυτές τις διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα λοιπόν να τα δούμε αυτά όταν δουλεύουμε πάνω στο κείμενο. Να βρούμε έναν τρόπο να υπάρχει ταυτόχρονη ενημέρωση από πλευρά σας. Σε σχέση με τον κύριο Πίπερ να σας πω ότι νιώθω μεγάλη ενθάρρυνση, γιατί Η οπτική γωνία που υιοθετεί είναι παρεμφερής με τη δικιά μου. Στόχος λοιπόν αυτής της ακρόασης και της αλληλοπίδρασης σήμερα δεν είναι βεβαίως να εξετάσουμε τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Ε, θα ολοκληρώσω κόπο εδώ, αλλά θα ήθελα να σχολιάσετε και εσείς τα λεγόμενά μου. Σίγουρα περιμένουμε από όλου να εργαστούν ικανοποιητικά για να έχουμε ένα στερεονομικό εργαλείο. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Κράμερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, τι πιστεύω εγώ. Όταν αρχίζουμε να δακτυλοδείχνουμε διαφόρους για τον αθέμητο διεθνή ανταγωνισμό, ε, να μην ξεχάσουμε ότι θα έχουμε τρία δάχτυλα που θα δείχνουν προς την Ευρώπη. Γιατί και στο εσωτερικό της Ευρώπης είναι αθέμητος ο ανταγωνισμός. Ένα στα δύο αεροδρόμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ελληματικό. Το δείχνουν τα στοιχεία έτσι στην Ευρώπη. Στη Γερμανία, αν κοιτάξουμε τι γίνεται, θα ήμουν χαρούμενος. Έχουμε 23 διεθνούς, διεθνείς στη Γερμανία, 17 είναι ελληματικοί. Δεν έχουμε λοιπόν θεμητό ανταγωνισμό καθόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δεν καταφέρνουμε να ρυθμίσουμε τα του οίκου μας, δεν μπορούμε να με ψημιρούμε ότι άλλοι ε, προχωρούν σε αθέμητο ανταγωνισμό. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και αεροδρόμια φτηνά και φτηνές αεροπορικές εταιρείες που είναι σχεδόν ε, δωρεάν η προσγείωση και απογείωση. Μετά έχουμε και κρατικές ενισχύσεις έμεσες, έτσι. Και νόμιμες έτσι κι αλλιώς, αλλά και έμεσες. 30 δισεκατομμύρια τους χαρίζει ο φορολογούμενος το χρόνο στις ε, αεροπορικές εταιρείες γιατί δεν πληρώνουν ΦΠΑ, δεν πληρώνουν κυρόζινη, τέλη, τα, τα ξέρετε, τα λέω συνέχεια, ενώ στο σιδηρόδρομο ισχύει αυτό. Ε, και ξέρω ότι υπάρχουν πολλές διαπραγματεύσεις για να ξεπεράσουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό και να συμφωνήσουμε με άλλες εταιρείες και με άλλα κράτη, αλλά αυτό κρατάει χρόνια και δεν καταλήγει πουθενά και δεν τα βρίσκουμε. Άρα μην σηκώνουμε και κουνάμε το δάχτυλο στους άλλου. Είχαμε πάει στον Καναδά με την Επιτροπή μα και ρωτήσαμε και μα είπαν ε, ότι όλοι οι αερολιμένε στον Καναδά είναι κερδοφόροι. Θα ήταν καταπληκτικό παράδειγμα για μα. αλλά απέχουμε πόρο. Και τι κάνουμε εκεί. Και όταν μας στιγματίζουν οι άλλοι ότι δεν κοιτάτε τα δικά σα που έρχεστε και μα κουνάτε το δάχτυλο. Γιατί εκεί πραγματικά θα βρεθούμε σε δινή θέση. Χρειάζεται σοβαρότητα εδώ, στοιχειώδες. Γιατί και τα τέλη αεροδρομή είναι πολύ διαφορετικά. Στη Φραγκφούρτη 40-50 ευρώ πληρώνεις για να προσγειωθείς και στο Αμβούργο 2-3 ευρώ, κάτι τέτοιο. Εκεί, εκεί δεν πρέπει να υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές για να μην επιδοτούν και να μην χρηματοδοτούν οι φορολογούμενοι. Ε, την αέρια κυκλοφορία γιατί ξέρουμε ότι οι εκπομπές εκεί ψηλά είναι τρεις ή τέσσερις φορές πιο επικίνδυνες ε, από ότι στο έδαφος. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κράμερ. Η κυρία Άγνοτσου. ευχαριστω πολυ ευχαριστω πολυ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Κορνέλης για την παρουσίασή σας. Δεν ε, θέλω να γίνω δυσάρεστη. Θέλω όμως εκ προημίου να πω ότι για να δώσει ένα τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον αθέμητο ανταγωνισμό θα έπρεπε να είχε δράσει πολύ νωρίτερα και μάλιστα ε, τον αθέμητο ανταγωνισμό τον δημιούργησε ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την παραδοσιακή πολιτική ε, της υπέρ ενός ανελαίτου ανταγωνισμού. Οι πρώην κρατικές ή εθνικές ε, αεροπορικές εταιρείες γονάτισαν και ε, τα κράτη έπρεπε ας πούμε να καθίσουμε στα βρωμένα χέρια να βλέπουν τις εταιρείε τους να καταραίουν σιγά σιγά γιατί δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις αεροπορικές εταιρείε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή τις χώρες του κόλπου γενικότερα οι οποίες όμως ε, εταιρείε ε, έχουν ένα σωρό ενισχύσεις από τα δικά τους κράτη και τις δικές τους κυβερνήσεις. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προστατεύσει αποτελεσματικά τον κλάδο. Καλώς. Αλλά γιατί δεν το κάνατε πιο πριν. Υπάρχει ο κανονισμός του 2004 που θέλετε να αντικαταστήσετε. Αλλά εδώ και 13 χρόνια δεν ισχύει. 13 ολόκληρα χρόνια οι εταιρείε μας έχουν υποστεί αθέμητο ανταγωνισμό χωρίς να έχουν μπορέσει να αντιδράσουν. Γιατί ο κανονισμός δεν ήταν καθόλου προσαρμοσμένος στις ανάγκες των αερομοτοφορών και δεν μπόρεσε και να λειτουργήσει ούτε να εφαρμοστεί. Τώρα ως προς αυτά που προτείνεται. Χαιρόμαστε γιατί υπάρχει κήρυξη ερευνητική διαδικασία. υπάρχουν εξελίξεις θετικέ σε σχέση με τον προηγούμενο κανονισμό για τον ε, ορισμό της τεκμηρίωσης που ε, δικαιολογεί την έναρξη της ε, διοικητικής εξέτασης της ΕΔΕ, ε, όταν δηλαδή ε, ε, υπάρχουν πρακτικές που μπορεί να πλήξουν τον, την εταιρεία και μπορεί να δώσουν λαβή για θέμη του ανταγωνισμού και το καθεξής. Η διαδικασία προσφυγής που προτείνεται πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν είναι νορμάλ και φυσιολογικό, μόνο ο κλάδος να μπορεί να προσφεύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να μην μπορούν, ούτε οι αερομεταφορείς να μπορούν, αλλά μόνο οι κατασκευαστές. Ωστόσο, κάποια στοιχεία θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Οι προθεσμίες έναρξης και λήξης μιας έρευνας θα πρέπει να είναι πολύ πιο ε, λίγες και μικρές για να είναι αποτρεπτικός ο κανονισμός. Και πρέπει να υπάρχουν και προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα όσο ε, ε, γίνεται έρευνα αλλά και μηχανισμός για να συμμορφωθούν τα μέρη με την τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε το σημείο Β του άρθρου 12, εδάφιο 2 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υιοθετεί μέτρα αποκατάστασης επανόρθωσης εάν αυτά είναι ενάντια των συμφερόντων της Ένωσης. Άρα, αν μια τρίτη χώρα ενδιαφέρεται, αρκεί να απειλήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εμπορικά αντίπεινα για να καταφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κλείσει αμέσως την έρευνα και να μην απαιτήσει τίποτα, ακόμα και να αποδεχθούν ε, ε, ε, στοιχεία θέμη του ανταγωνισμού. Πώς θα την εφαρμόσετε αυτή την απόφαση και πώς θα την δράσετε ε, σε αυτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν αντίπεινα ως μέτρα από τις τρίτες χώρες οι οποίες θα τεθούν στο στόχαστρο μιας διαρευνητικής διαδικασίας καθόλου τεκμηριωμένης. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπλουμ, ε, Κλουμ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για την πολύ σαφή σας παρουσίαση. Με ενθαρρύνουν τα λόγια σας. Λέτε ότι ο κανονισμός είναι, έχει ως σκοπό να διασφαλίσει τον ανταγωνισμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι διαφάνειες που δείξατε τονίσαν τη διασύνδεση, τη συνδεσιμότητα, πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Έχουμε εμπορικέ συμφωνίες με την Ιαπωνία, με το Καναδά, με τη Σιγκαπούρη, με την Αυστραλία, ο Σονούπο, Επομένως η διεθνή συνδεσιμότητα είναι πολύ σημαντική και για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Συμφωνώ απολύτως. Πράγματι, χρειαζόμαστε κάτι για να αντικαταστήσουμε τον προηγούμενο κανονισμό που δεν ήταν αρκετός και δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Είναι πολύ ενθαρρυντικά τα λόγια σας. Δίκαιη προσέγγιση, προστασία καταναλωτών και επιχειρήσεων ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες θα έχουν μια δίκαιη και σωστή προσέγγιση όπως και οι υπόλοιπες. Όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι συμφωνίες υφιστάμενες θα πρημοδοτηθούν, ειδικά οι συμφωνίες που έχουν εσωτερικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών και θα εξαντληθούν όλα αυτά τα εσωτερικά μέσα για την επίλυση των διαφορών. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ήδη υπάρχουν μηχανισμοί επίλυσης διαφορών στις συμφωνίες που έχουν ήδη συναυθεί σε αυτό το πεδίο. Συνοπτικά λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει ένα εργαλείο για να διαχειριστεί όλες αυτές τις προσφυγές. ακούμε διάφορα επιχειρήματα υπέρ των μεν και των δε. Ε, ε, δεχόμαστε διάφορα έγγραφα που δείχνουν ότι ο αερομεταφορέας έχει αθέμητες ενισχύσεις, επιδοτήσεις, κάποιους άλλους όχι. Ε, το σημαντικό είναι ότι έχουμε μια δομή, θα έχουμε μια δομή για να μπορέσουν όλα αυτά να κριθούν και να εξεταστούν σωστά. Από την παρουσίασή σας φαίνεται ότι η προσέγγιση σας είναι δίκη, είναι ισόρροπη, ισορροπημένη και με χαρά θα συνεργαστώ για την προώθηση αυτής της νομοθεσίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η λέξη κλειδί είναι ισορροπία προς όφελος των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και του διεθνούς εμπορίου. Ευχαριστούμε την κυρία Κλούν. Κύριε Κορνέλη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Δείξατε ότι ο ανταγωνισμός οξύνεται μεταξύ των διαφόρων ε, αερομεταφορέων. Και αυτό είναι περίεργο γιατί ξέρουμε ότι οι συνθήκες αυτές του ανταγωνισμού δεν ρυθμίζονται διεθνώς από κανένα νομοθετικό εργαλείο και αυτό είναι πολύ περίπλοκο. Επομένως, πώς θα τα καταφέρετε να πείσετε τις χώρες και μάλιστα τις χώρες μέλη που σήμερα είναι διάκειται εχθρικός ως προς την ιδέα αναθεώρησης του κανονισμού. Αυτό είναι και το πρώτο στάδιο. Κάποια κράτη-μέλη θεωρούν ότι αυτός ο κανονισμός μοιάζει με προστατευτισμό και το καθεξής και άρα είναι πολύ δύσκολο να δεχθούν επανεξέτασή του. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Μηχανισμός προστασίας. Δεν είναι πολύ σαφής. Δεν είναι σαφή αυτά που λέτε. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Τι εννοείται με τα λόγια σας μηχανισμός προστασίας. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Και τέλος. Θα ήθελα να ξέρω κάτι σε σχέση με τα μέτρα αποζημίωσης ή αποκατάστασης, ειδικότερα μεταξύ των διεθνών μεταφορών στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών. Υπάρχουν διάφοροι φόβοι. Πώς θα τα επαναπροσδιορίσουμε όλα αυτά. Από ό,τι φαίνεται πήρα το λόγο ως πρόεδρος, ενώ είχαμε άλλους στην αίθουσα ομιλητές που ήθελαν να πάρουν το λόγο. Παρακαλώ. Δεν ε, σας έχω στον κατάλογο ομιλητών, σας προσθέτω όμως. Ο κύριος Βαν Μίτελμπεργκ και η κυρία Ντεμόντ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν κάνετε εσεί τόσε ενδιαφέρουσε ερωτήσει, θα περιμένω τη σειρά μου να πω και εγώ δύο λόγια. Ε, καλωσορίζω πρώτα απ' όλα την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί σε διάφορα ψηφίσματά του το Κοινοβούλιο είχε καταστήσει σαφές πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ε, θεμητό ανταγωνισμό και μάλιστα με συγκρίσιμα στοιχεία και μετρήσιμα μεταξύ των διαφόρων αερομεταφορέων. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια σωστή απάντηση για να εξασφαλίζουμε ότι υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός. Και εγώ που είμαι και μέλος των φιλελευθέρων εδώ, καλωσορίζω κάθε είδους ε, πρωτοβουλία που τα βελτιώνει. Έχω και κάποιες ερωτήσεις όμως, γιατί στην πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρθηκε σε κάτι που στρέφεται κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και παραθέτω άρθρο 3, άρθρο 10, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να μην εκκινήσει μια διαδικασία διερεύνηση σε περίπτωση που τα αποτελέσματα και τα πορίσματα στρέφονται κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν στο, στο άρθρο 3 και στο άρθρο 10 περίπου τα ίδια αναφέρει για μέτρα αντισταθμιστικά και επανορθωτικά αλλά μπορεί να παραλείψει να το κάνει αυτό όταν στρέφεται κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό παρακαλώ πώς ορίζεται το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί μιλάμε για κανονισμό εδώ. Θα πρέπει να είναι λοιπόν και απέναντι ε, στο δικαστήριο αυτό ε, αδιάβροχο και ε, σύμπαγες. Ποιος το αποφασίζει λοιπόν, τα επαναρθωτικά μέτρα κτλ. Εάν το ε, προσβάλλει ένα αερομεταφορέ μιας τρίτης χώρας. Πώ ορίζεται λοιπόν το συμφέρον της Ένωσης. Είναι στο άρθρο 10, 2β. Επίσης, οι ρήτρε θεμητού ανταγωνισμού σε συμφωνίες ταυσιπλοίες. Υπάρχουν οι διεθνεί κανόνε. αυτό είναι το ένα πρώτο επίπεδο, ένα πρώτο στρώμα και σε περίπτωση που αυτές παραβιάζονται, ε, τι γίνεται σε δεύτερη φάση. Πώς έχει δυναμική. Γιατί τώρα διαπραγματεύεστε με τρίτες χώρες. Πώς αντιδρούν οι τρίτες χώρες στις διαπραγματεύσεις αυτές. Γνωρίζω πλήρως και απολύτως ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ε, εμπιστευτικέ, αλλά μήπως κάποια γενικότερα σχόλια να μας κάνετε. Και ακόμα μια ερώτηση. Μιλήσατε για το άρθρο 13 οικονομικές ε, υποχρεώσεις, επαναστατικά μέτρα κτλ. Ξέρουμε ότι σε διμερή βάση έχουμε μέτρα. Τι είναι οικονομικές επιβαρύνσεις και τι είναι κάθε μέτρο ισοδύναμης ή μικρότερης αξίας. Μπορείτε να μας δώσετε τρία παραδείγματα. Κατά την άποψή σας τι σημαίνει κάθε μέτρο ισοδύναμη ή μικρότερης αξίας. Και οι τελευταίε ερωτήσει μου έχουν να κάνουν με τα κράτη-μέλη. Γιατί ξέρετε ότι έγινε μια πρώτη συζήτηση, ένα γύρο τραπέζι στο Συμβούλιο με τα κράτη-μέλη. Αν δεν απατώ με τον Ιούνιο, υπάρχουν κάποιε επιφυλάξει, ιδιαίτερα από πλευρά των Βρετανών συναδελφών, εξ όσων κατάλαβα. Ίσως μετά το Brexit θα το λύσουμε και αυτό. Αλλά έχω την εξή ερώτηση. Εσείς τι μπορείτε να κάνετε, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρξει λίγο μεγαλύτερος ενθουσιασμός στις τάξεις των κρατών μελών στο Συμβούλιο. Πώς θα τους κινητοποιήσουμε για να λάβουν κάποια δράση, για να μας υποστηρίξει το Συμβούλιο, γιατί είναι κρίσιμος αυτός ο κανονισμός. Βέβαια, κάθε θεσμικό όργανο έχει το δικό του ρόλο να διαδραματίσει, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω πρέπει να είναι πολύ πιστική ιδιαίτερα για τα κράτη-μέλη που ε, έχουν τις επιφυλάξεις τους και τις αντιστάσεις τους για το κανονισμό 868 του 2004 και την αναθεώρησή του. Στην παρουσίασή σας είπατε ότι έχουμε τον ΠΟΕ, ας πούμε, για τον θεμητό ανταγωνισμό, αλλά τελικά θα πρέπει να εργαστούμε έτσι ώστε οι υπηρεσίες ε, αεροπόρων μεταφορών να ενταχθούν στον ΠΟΕ γιατί είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσω στους ψηφοφόρους ότι Boeing και η Airbus ε, μπορούν να υπάγονται στον ΠΟΕ, αλλά οι αερομεταφορείς όχι. Ξέρουμε τις ευαισθησίες που υπάρχουν και τις κατανοώ και εγώ. Από την άλλη όμως Υπάρχει μια έκφραση στα Ολλανδικά που λέει και που είναι ορίζοντα, δηλαδή προ τα πού το πάμε, πού θα καταλήξουμε, πού θέλουμε να φτάσουμε, ποια θα είναι η τελική ε, διευθέτηση των θεμάτων του ε, δίκαιου ανταγωνισμού και του θεμητού. Για μένα είναι ο ΠΟΕ. Πώ αντιδράτε σε αυτό, πώ τους βλέπετε, είναι το πρώτο βήμα προ την κατεύθυνση αυτή και τι θα πρέπει να κάνουμε για να πείσουμε τα κράτη-μέλη που διστάζουν ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Βαν Μίλτενμπουργκ, η κυρία Ντεμόντι έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σα ευχαριστήσω για την παρουσίαση αυτή. Θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση και μια ερώτηση. Παρατήρηση πρώτα. Το ζήτημα τη ευελιξία. Μα είπατε πολύ σωστά ότι θα πρέπει να υπάρχουν τιμωρητικά μέτρα, ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και τα ωφέλη που ενδεχομένω να υφίστανται, όσον αφορά τις παρεχόμενες αυτές αεροπορικές υπηρεσίες. Μας δώσετε όμως και κάποια δεδομένα και φάνηκε ότι διπλασιάστηκε ο ρυθμός των καθημερινών πτήσεων από το 1992 στο 2016 και μεμορίζει το 2050. Ξέρουμε ότι θα υπάρξει επίσης μια ακόμα σημαντικότερη αύξηση της ενέργειας κυκλοφορίας. Άρα μιλάμε για πραγματική κυκλοφοριακή συμφόρηση στους ευρωπαϊκούς ουρανούς, άρα πρέπει να παρέχουμε όσο δυνατόν πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες προκειμένου να μπορούμε να εξυπηρετούμε πραγματικά τους πολίτες και να μπορούν να έρχονται και λίγο πιο κοντά. Αλλά μην ξεχνάμε και την ανάπτυξη την περιφερειακή. Αν δεν υπάρχει η απαραίτητη αεροπορική μεταφορά, η σχετική δηλαδή υπηρεσία που να παρέχεται από τον κλάδο αυτό, τότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κάποιοι προορισμοί οι οποίοι να μην εξυπηρετούνται καθόλου, γιατί μπορεί να μην θεωρηθούν καν τουριστικοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν κάποιοι προορισμοί στους οποίους να μπορεί να πηγαίνει κανεί με χαμηλού ναύλου τελικά, γιατί αυτό θα συμβάλλει πάρα πολύ στην οικονομική τη ανάπτυξη. Θεωρώ λοιπόν ότι βρίσκεστε στη σωστή κατεύθυνση, ιδίως όσον αφορά τις εξόχως απόκεντρε περιοχές. Από την όμως έχω και μια ερώτηση. Όσον αφορά την εφαρμογή αυτού του κανονισμού σε σχέση με τις συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Εγώ είμαι η συγγήτρια για τις συμφωνίες που έχουμε με τις χώρες του κόλπου αλλά αυτό αφορά βασικά και όλες τις τρίτες χώρες και όχι μόνο αυτές τις χώρες του Περσικού κόλπου. Πώς θα εφαρμόζεται ακριβώς αυτός ο κανονισμός, θα υπερισχύει τελικά η συμφωνία όσον αφορά το ζήτημα του ανταγωνισμού ή θα υπερτερεί τελικά ο κανονισμός. Ξέρετε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε περίπτωση παραβίαση των εφαρμοστέων διεθνών υποχρεώσεων ή σε περίπτωση πρακτικών που εισάγουν διακριτική μεταχείριση, ποιο από τα δύο τελικά θα ισχύει, η συμφωνία που έχουμε συγγράψει με τη χή χώρα ή ο κανονισμό. Σα ευχαριστούμε κυρία Ντεμόντε. Να ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Κορνέλη τώρα, προκειμένου να μα διαφωτίσει σχετικά με όλε αυτέ τι ερωτήσει. Έχετε το λόγο. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πίπερ και γενικότερα τους κοιόδης συγητές που δείξαν τέτοιο ενδιαφέρον για την πρόταση αυτή και προφανώς προσβλέπω για περαιτέρω συνεργασία με εσά και όλη η ομάδα μου, όλοι μου οι συνεργάτες στην διαθεσή σας προκειμένου να σας δώσουν περισσότερα στοιχεία εφόσον τα χρειάζεστε. Σας ευχαριστώ επίσης πολύ για την γενικότερη και ευρύτερη υποστήριξη που δείχνετε προς την πρόταση αυτή κανονισμού. Βλέπω ότι πολλοί αν όχι όλοι θεωρείται ότι είναι μια ισόρροπη και αναγκαία πρόταση. Αυτό είναι ιδιαίτερα θαρρυντικό για μένα. Βέβαια, ορισμένοι είπατε ότι υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις τις οποίες θα πρέπει να τονίσουμε λίγο περισσότερο ή που θα πρέπει να προσθεθούν στην πρόταση κανονισμού. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο. Τώρα, ας επανέλθω σε κάποιες σημαντικές συγκεκριμένες με παρατηρήσεις που γίνανε. Ο κύριος Τελίτσκα αναφέρθηκε στην αξιολόγηση αντικτύπου και στο ζήτημα της συνδεσιμότητας. Προφανώ η αξιολόγηση αντικτύπου, η αξιολόγηση επιπτώσεων και η διεξαγωγή μια αξιολόγηση είναι δύσκολο έργο, μην το ξεχνάμε αυτό και καθίσταται ακόμα πιο δύσκολο όταν μιλάμε για το πεδίο αυτό που ουσιαστικά είναι ένας κανονισμός πλαίσιο, ένας κανονισμός που δημιουργεί μια διαδικασία. Θέτει κριτήρια, θεσπίζει μια διαδικασία, δεν υπησέρχεται όμως σε πραγματικές περιπτώσεις και όπως το είπατε πολλοί από εσά σωστά, ο βασικό μα στόχο και προτού τεθεί σε ισχύ ο κανονισμό αυτό είναι να δούμε και να αξιολογήσουμε συγκεκριμένε περιπτώσει και καταστάσει. Είναι δύσκολο λοιπόν να αποτιμήσουμε αριθμητικά ή ποσοτικά ποιο θα είναι ο αντίκτυπο του κανονισμού αυτού για περιπτώσει περιπτώσεις οποίε δεν τις γνωρίζουμε ακόμα. Τούτων λεχθέντων θεωρώ ότι, μολονότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι περιορισμοί, καταφέραμε παρόλα αυτά να κάνουμε μία πιστική αξιολόγηση επιπτώσεων και λέω πιστική γιατί ουσιαστικά απαντά τα πιο βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει οι εξολόγηση ε, επιπτώσεων, που είναι ή κάνουμε κάτι ή δεν κάνουμε τίποτα. Ή αν θα πρέπει τελικά να λάβουμε δράση σε διεθνές επίπεδο με τον ΠΟΕ και τον ΙΚΑΟ ή αν θα πρέπει να περιοριστούμε σε ευρωπαϊκά μόνο μέσα και εργαλεία. Όπως το είπαμε και εμείς και το είπατε και εσείς, οι περισσότεροι από εσά θεωρούμε ότι ένα συνδυασμό και των δύο είναι το ευκταίο. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει και σε διεθνέ επίπεδο να λάβουμε δράση με τον ΠΟΕ και τον ΙΚΑΟ, αλλά και σε διμερές επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τι αδυναμίε λοιπόν αυτέ και του περιορισμού αυτού που μπορεί να υπάρχουν σε πολλά συγκεκριμένα σημεία, παρόλα αυτά θεωρώ ότι καταλήξαμε σε πολύ καλά συμπεράσματα στα πλαίσια αυτή τη εξολόγηση επιπτώσεων και τα οποία ενέκριναν και ε, ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Τώρα το ζήτημα της ενδεσιμότητας. Αυτό έχει αποτελέσει ανησυχία και για εσάς αλλά και για το Συμβούλιο και γι' αυτό το λόγο το έθιξα τόσο πολύ στα πλαίσια της παρουσίασής μου. Η συνδεσιμότητα είναι το σημείο θετηρίας για μας. Σε καμία περίπτωση δεν είναι το θύμα του κανονισμού αυτού. Είναι μάλλον αυτό το οποίο προωθούμε μέσω αυτής της πρώτης κανονισμού. Αυτή είναι η οπτική μας γωνία. Χρειαζόμαστε ως το δυνατόν περισσότερου παίκτες, περισσότερου φορείς που δραστηριοποιούνται σε μια πραγματικά ανταγωνιστική αγορά. Δηλαδή μια αγορά όπου δεν θα υπάρχει διακριτική μεταχείριση, αλλά που θα είναι απόλυτα ανοιχτή. Ο κανονισμό λοιπόν αυτό μπορεί να μα βοηθήσει να το κάνουμε αυτό εκεί που δεν έχουμε άμεση δικαιοδοσία, δηλαδή στο εξωτερικό, εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, ακόμα και ο κανονισμό αυτό ε, έχει ω στόχο να μα βοηθήσει εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, εμεί ε, αυτό το οποίο προτιμούμε ω διαδικασία και παντώ τώρα σε μια άλλη ερώτηση είναι οι διμερεί σχέσει και ουσιαστικά οι λύσει που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευση. Το μέσο αυτό το οποίο σας προτείνουμε εδώ πέρα θα χρησιμοποιηθεί όταν δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί άλλη διαδικασία, όταν δεν μπορούμε να συνεργαστούμε στα πλαίσια μια συμφωνία. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν πρόκειται εμεί να χρησιμοποιήσουμε άμεσα το μέσο αυτό. Πρώτα θα κάνουμε συζητήσει, πρώτα θα κάνουμε πραγματεύσει, είτε εμεί είτε τα κράτη-μέλη με τι τρίτε χώρε, αλλά δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να φτάσουμε στα διέξοδο και τότε δεν θα έπρεπε να μένουμε χωρίς κανένα άλλο διαθέσιμο μέσο ή εργαλείο, γιατί στην περίπτωση αυτή όντως κινδυνεύει να ζημιωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε, αυτή είναι η σειρά που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Καταρχάς, η διεθνείς που θελουμε να ακολουθησουμε καταρχας οι διεθνεις κανονες και απαντώντας και στο ερώτημά σας θα εξακολουθούμε να προωθούμε τους κανόνες αυτούς, ιδίως στα πλαίσια του ΙΚΑΟ, Βέβαια πρέπει να πω ότι εμείς εδώ οι Ευρωπαίοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία προωθεί περισσότερο την ανάγκη διεθνών κανόνων και λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες που να ισχύουν διεθνώς. Υπάρχουν άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν το επιθυμούν αυτό καθόλου. Ακόμα και χώρες που γενικά λένε ότι είναι υπέρ των ανταγωνιστικών αγορών όπως οι ΗΠΑ. Όταν μιλάμε για την αεροπορία με τις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ διστακτικές όταν πρέπει να θεσπίσουμε διεθνείς κανόνες και έπειτα έχουμε και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και εκεί θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση, αλλά δεν είναι πολύ ρεαλιστικό να ελπίσουμε ότι μέσα στα επόμενα δύο-τρία χρόνια θα έχουμε εκεί πέρα ένα αποτελεσματικό διεθνές εργαλείο. Ο κύριο Κράμερ στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ζήτημα του ανταγωνισμού στο πλαίσιο τώρα εντό Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό αποτελεί για μα εξίσου σημαντική ανησυχία. Και όπω είπα και στην αρχή τη παρέμβασή μου, θα θέλαμε η προσέγγιση μας να θεωρηθεί ως μια ολιστική προσέγγιση. Στα πλαίσια της στρατηγικής για την αεροπορία έχουμε προωθήσει διάφορες πρωτοβουλίε. Μία από αυτές είναι και αυτή που σας παρουσίασα σήμερα όσον αφορά τους αερολιμένε και τη μεταξύ αυτών, το μεταξύ αυτών ανταγωνισμό. Προφανώς εμείς δεν θέλουμε να έχουμε αεροδρόμια, αερολιμένε για του οποίου δεν υφίσταται κάποια αγορά. Η Επίτροπο Μπούλτ το έχει πει αυτό πολλέ φορέ Και έχουμε και πολύ αυστηρού κανόνε όσον αφορά τι κρατικέ ενισχύσει προ αερολιμένες ή όσον αφορά τις επενδύσεις ή την επενδυτική αερογή προς τα αεροδρόμια αυτά. Και σε καμία περίπτωση βέβαια θα πρέπει να προβλέπετε στα πλαίσια των κοινοτικών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις να καλύπτονται ποτέ τα ελληματικά αεροδρόμια, οι ελληματικοί αερολιμένες. Και πάλι εγώ θεωρώ ότι σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου έχουμε πολύ ανταγωνιστικούς αερολιμένες. Πολλές φορές τα τέλη διαφέρουν από τον ένα ρολιμένα στον άλλον, όντω, αλλά αντικατοπτρίζουν σε κάθε περίπτωση τι διαφορέ που υπάρχουν όσον αφορά το κόστο, το επενδυτικό, τι διαφορέ στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και βέβαια τα τέλη αυτά, όπως ξέρετε, θεσπίζονται βάσει των κανόνων που υπάρχουν στην σχετική οδηγία για τα τέλη αεροδρομίου. Άρα θα πρέπει και αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας κάθε φορά που συγκρίνουμε τα αεροδρόμια μεταξύ τους. Μπορεί να έχουμε για παράδειγμα ένα αεροδρόμιο το οποίο επεκτείνεται, το οποίο προβλέπει, θα χτίσει, θα δημιουργήσει νέους αεροδιαδρόμους ή νέες υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή είναι λογικό τα τέλη να είναι υψηλότερα γιατί ακριβώς χρηματοδοτούν τις νέες αυτές επενδύσεις. Πάντως θα αρχίσουμε να αναθεωρούμε και την υπηρεσία για τις υπηρεσίες, την 1008, αλλά και την υπηρεσία που έχουμε για τα τέλη, την οδηγία με που έχουμε για τα τέλη αεροδρομίου. Επομένως βλέπετε ότι όλες οι πτυχές τελικά του κανονισμού αυτοκλησίου θα αναθεωρηθούν μέσα στα επόμενα έτη. Και βέβαια θα έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουμε σε όλα αυτά τα ζητήματα. Η κυρία Αρνοτού αναφέρθηκε στη συνέχεια στο ζήτημα του χρονοδιαγράμματος ε, και το αν θα ήταν δυνατόν να έχουμε κάποια προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα. Ξέρετε, μπορούμε όντως να κινηθούμε γρήγορα Τίποτα δεν μα εμποδίζει και γι' αυτό το λόγο υπάρχει η έννοια όχι μόνο τη ζημία αλλά και τη απειλή ζημία. Δηλαδή μπορούμε να αναλάβουμε δράση ακόμα και δεν έχει λάβει χώρα ζημία και είμαστε απλώ πεπισμένοι και σίγουροι ότι αυτή θα λάβει χώρα κάποια στιγμή στο μέλλον. Αρκεί να υπάρχει λοιπόν απειλή ζημία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αναλάβει γρήγορα δράση όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τώρα, το ζήτημα της, του συμφέροντος Ευρωπαϊκής Ένωση, Αυτό το θίξανε πολλοί ευρωβουλευτές. Κοιτάξτε, είναι όντω κεντρικό σημείο τη πρόταση ε, κανονισμού και θα αποτελέσει σημαντικό σημείο συζήτηση και στο Συμβούλιο πώ μπορούμε να ορίσουμε το συμφέρον τη Ένωση. Εμεί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει έννοια αυτή, δεν την επινοήσαμε εμεί, υφίσταται ήδη σε όλα τα υπόλοιπα μέτρα προστασία του εμπορίου. Δεν θα πρέπει ουσιαστικά, θα πρέπει να αποφύγουμε την κατάσταση εκείνη όπου κάποιο καταθέτει μία καταγγελία ξεκινάει μετά μια διαδικασία την οποία δεν μπορούμε τίποτα να αναχαιτήσουμε και η οποία τελικά οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα το οποίο στρέφεται κατά του ίδιου του συμφέροντος των Ευρωπαίων πολιτών. Λέμε λοιπόν ότι κάποια στιγμή στην αρχή της όλης διαδικασίας θα πρέπει να έχουμε μία γενικότερη, πιο σφαιρική αντιμετώπιση της κατάστασης και να δούμε τελικά αν αξίζει να αναλάβουμε δράση ή όχι. Για παράδειγμα, από τον κανονισμό για την προστασία του εμπορίου ή, για τις, ή στα πλαίσια των διαδικασιών dumping που έχουμε, πολλές φορές βλέπουμε ότι προσπαθούμε να εξορροπήσουμε συμφέροντα παραγωγών και καταναλωτών. Και βάσει αυτών έχουμε αποφασίσει πολλές φορές ότι τελικά αξίζει ή ότι τελικά δεν θα έπρεπε να επιβληθούν κάποια μέτρα. Είναι δύσκολο να γίνει κανεί πιο συγκεκριμένο στο κείμενο αυτό κάθε φορά που αναφερόμαστε στο συμφέρον τη Ένωση. Γιατί αν γινόμασταν πιο συγκεκριμένοι και πιο περιοριστικοί, τότε αυτό θα ήταν αντιπαραγωγικό. Δεν θα μα επέτρεπε, τελικά ο κανονισμό να δούμε την πιο σφαιρική εικόνα. Όντω υπάρχουν, μάλλον δεν υπάρχουν μέτρα τα οποία να είναι πιο συγκεκριμένα ούτε στου άλλου κανονισμού. Τώρα το ζήτημα τη συζήτηση στο Συμβούλιο. Το ακούσατε πολύ σωστά ότι όντω δίστανται οι απόψεις μεταξύ των κρατών μελών. Η δική μας εντύπωση είναι ότι αυτό οφείλεται στο ότι έχουν παγιωθεί ήδη κάποιες απόψεις προτού καν υποβληθεί η πρόταση αυτή κανονισμού, που έχει να κάνει αυτό με μονομένες προσδοκίες που έχουν κάποια κράτη-μέλη. Προσπαθούμε να σημειώσουμε αυτή τη στιγμή πρόοδο, λέγοντα ότι α ξεχάσουμε λίγο τα δημοσιεύματα στον τύπο που διαβάσαμε πέρυσι και α δούμε τελικά πραγματικά τι λέει το κείμενο αυτό και τι προβλέπει τελικά προκειμένου να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμό. Προκειμένου να μην συμβούν αυτά τα οποία φοβάται ότι μπορούν να συμβούν ένα κράτο μέλο. Ότι δεν θα κλείσουμε δηλαδή όλες τις πτήσεις ή τις διασυνδέσεις αεροδρομίου με μια χώρα που εμπλέκεται σε μια καταγγελία, για παράδειγμα. Προφανώς δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πολλές ε, ρήτρε διασφάλιση ήδη στο κείμενο και αυτό προσπαθούμε να πούμε στα κράτη-μέλη και νομίζω ότι εδώ εσεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχετε ήδη δει αυτό. Ελπίζω λοιπόν ότι και το γενικότερο κλίμα και η γενικότερη εντύπωση αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο θα εξελιχθεί, ότι να αρχίσουν τα κράτη-μέλη σιγά σιγά να καταλαβαίνουν περισσότερο τι θέλουμε να πετύχουμε με το νέο αυτό μέσο. Και βέβαια προσβλέπουμε και στη διοργανική συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, η οποία ελπίζω ότι θα είναι ιδιαίτερα θετική. Τώρα, οι διμερείς συμφωνίες ή οι εντιμερεί συμφωνίες που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Ως προς αυτό πρέπει να σας πω ότι μα έχουν δοθεί θετικές απόψεις από τις χώρες εκείνες με τις οποίες διαπραγματευόμαστε, γιατί και αυτές οι τρίτες χώρες θεωρούν ότι η πρόταση αυτή είναι ισορροπημένη, βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και περιστατικά, ότι όντως σέβεται το δικαίωμα υπεράσπισης και ότι δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, όλα αυτά που φοβόμασταν θα αποτελούσαν τελικά ανησυχίε για κάποια κράτη-μέλη, αυτά που είχαν προβληθεί ω αδύναμα σημεία αυτή τη πρόταση, τελικά δεν έχουν γίνει αντιληπτά κατά αυτόν τον τρόπο από τρίτε χώρε που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσει που έχουν συνάψει συμφωνίε με κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπω σα είπα, είμαστε υπέρ των διαπραγματεύσεων και προφανώ θέλουμε να προωθήσουμε τι εταιρικέ αυτέ σχέσει, οι οποίε όντω θα περιέχουν πολύ συγκεκριμένε λεπτομερεί ρήτρε για το πώς μπορούμε επιχειρηματικά να δραστηριοποιούμεθα στις χώρες αυτές και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τελικά τα συμφέροντα των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χάρη στις οποίες τελικά ρήτρες δεν θα χρειαστεί πιστεύω καν να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον κανονισμό. Μου ζητήσατε να σας δώσω κάποια παραδείγματα για ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν πέρα από τα πρόστιμα. Κοιτάξτε, οποιοδήποτε μέτρο θα μπορούσε να ληφθεί που έχει να κάνει με αεροπορικέ μεταφορέ, αεροπορικέ υπηρεσίε, πρόσβαση σε αεροδρόμια, πρόσβαση σε χρονοθυρίδε, χρησιμοποίηση άλλων υπηρεσιών που απαιτούνται για την παροχή αεροπορικών μεταφορών. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όλα τα επιχειρησιακά αυτά μέτρα είναι πιθανά πέραν αυτών που θα οδηγούσαν ή εμάς ή τα κράτη-μέλη σε μία παραβίαση διεθνών διμερών συμφωνιών. Τέτοια μέτρα προφανώς σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ληφθούν. Στην πράξη και ήδη προβλέπεται στον κανονισμό που έχει να κάνει με τις χρονοθυρίδες, με λιγότερο όμως περίπλοκο τρόπο, ότι αν ένα αεροδρόμιο τρίτης χώρας εισάγει διακρίσεις κατά ευρωπαϊκών ε, αεροπορικών εταιριών και δεν μας δίνει χρονοθυρίδες, έτσι μπορούμε και εμείς να προχωρήσουμε σε αντίστοιχα μέτρα, περιορίζοντας τις χρονοθυρίδες για τους αερομεταφορείς από την τρίτη αυτή χώρα. Και μάλιστα αυτό έχει προκύψει πριν από κάποια χρόνια. Χρησιμοποίησαμε το μέτρο αυτό και η διακριτική μεταχείριση μέσα σε λίγες μόνο ώρες, μέσα σε λίγα 24 ώρα, αποσύρθηκε. Επομένω βλέπετε ότι όντως τα μέτρα αυτά έχουν έναν αποτρεπτικό χαρακτήρα. Για τον ΠΟΕ απάντησα ήδη και τα όσα είπε η κυρία Ντεμόντε για την περιφερειακή ανάπτυξη, τι βλέπουμε, ότι η ίδια η εσωτερική αγορά οδήγησε σε τεράστια αύξηση των ε, δρομολογίων. Είναι τριπλάσια από ό,τι στην αρχή της εσωτερικής αγοράς όταν πρώτο δημιουργήθηκε. Δηλαδή πολλές πόλεις που στο παρελθόν δεν είχαν αεροπορική σύνδεση, τώρα αυξάνεται και έχουμε περισσότερες περιφερειακές ε, συνδέσεις και δρομολόγια με απευθείας πτήσεις και όχι ανταποκρίσεις μέσω μεγάλων κόμβων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ε, έχουμε τη δυνατότητα να υποχρεώσουμε για καθολική υπηρεσία ε, υπηρεσία δημοσίου συμφέροντος και τον Ιούνιο, γιατί είδαμε ότι οι χώρες διστάζουν να καταφύγουν σε αυτό και πώς και γίνεται και πότε επιτρέπεται κτλ. Αυτά. Νομίζω ότι κάλυψα τα βασικά σημεία, Πρόεδρε. Merci Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κορνέλης. Πραγματικά προσπαθήσατε να φωτίσετε κάποια σημεία που μας απασχολούσαν κάποιες σκιές που είχαμε για τον κανονισμό αυτό. Πρώτη φορά ε, συζητούμε το θέμα αυτό μαζί σας και να είστε βέβαιος ότι θα σας ξανακαλέσουμε όσες φορές χρειάζεται. Μπορείτε να ε, υπολογίζετε στη δική μου βοήθεια ακριβώς έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και είστε πάντα ευπρόσδεκτος στην Επιτροπή μου. Et maintenant, λοιπόν, συνεχίζει τη συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών. Άρα θα ζητήσω μια σύντομη διακοπή για να σταματήσει το web streaming και να μπορέσει το κοινό να αποχωρήσει έτσι ώστε να συνεχίσουμε και κλεισμένο των θυρών. Παρουσία των βουλευτών για το επόμενο θέμα. Δύο λεπτά έχετε για να βγείτε από την αίθουσα.